Κύριε έχετε το λόγο. Ευχαριστώ για την εμπιστοσύνη που μου δείξατε στα πλαίσια αυτής της εργασίας για, την, ε, θέμα της ανάπτυξης και ζήτησα το λόγο για να σας ζητήσω να γίνουν τα πάντα ούτως ώστε ε, να περάσει το Σεπτέμβριο στην Ολομέλεια του Στρασβούργου. Αυτό θα επιθυμούσα. Πρόεδρος, καλώς. Έχει ήδη προβλεφθεί κάτι τέτοιο. Ε, υπάρχει το πρόγραμμα το προσωρινό. Πρόεδρος, θα πρέπει φυσικά ο καθένας να κάνει το, το αρμόζον λόμπινγκ στην ε, πολιτική του ομάδα. Τώρα συνεχίζουμε για το προπολογισμό της Ευρωπαϊκής Ένωσης για το 2013, το γενικό προπολογισμό. 27 Μαρτίου και 14 Μαΐου είχαμε τη δυνατότητα να ανταλλάξουμε κάποιες ε, απόψεις σε σχέση με τις προτεραιότητες μας. Τώρα έφτασε το σημείο να, θα λέγαμε να περάσουμε στην πράξη όσον αφορά τις προτεραιότητες μας, να κάνουμε συγκεκριμένες προτάσεις για αυτό το σχέδιο προπολογισμού. Οι συγητές μας για αυτό το 2013 είναι ο Γκέι Μίτσελ. Μας έκανε μια ανακοίνωση και ανέφερε ότι έχει τροπολογίες, τις οποίες έχετε στο φάκελό σας. Όπως ξέρετε, η Επιτροπή Προπολογισμών εν ονόμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου θα κάνει διαπραγματεύσεις με το Συμβούλιο. Η γνωμοδότησή μας θα είναι η συμβολή που έχουμε να κάνουμε εμείς και είναι σημαντική σε σχέση με το τμήμα του προβλησμού που έχει να κάνει με τις δικές μας αρμοδιότητες θα κάνουμε τα πάντα για να πείσουμε τους συναδέλφους μας στην Επιτροπή Προπολογισμών, ούτω ώστε να είναι υπέρ των προτάσεών μας και να λάβουν ναι, υπόψη τη δική μας θέση για τη συνέχεια της διαδικασίας. Ο Γκέι Μίτσελ, που είναι και εισηγητής μας, του θα αναλάβει τώρα το λόγο, θα λάβει το λόγο για να κάνει την παρουσίαση των ε, γενικών ε, κατευθυντήρων γραμμών μας. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Θέλω καταρχήν να πω ότι η πρώτη σειρά τροπολογιών μου το έγγραφο που κυκλοφόρησε την προηγούμενη εβδομάδα περιλαμβάνει τις, τις προτάσεις Κομισιόν για το σχέδιο προϋπολογισμού του 2013 και τις συγκεκριμένες γραμμές του υπολογισμού που ε, θέλαμε να προωθήσουμε. Την προηγούμενη εβδομάδα το Συμβούλιο έδωσε συγκεκριμένα νούμερα για τη θέση του στο σχέδιο προϋπολογισμού και αυτά κυκλοφόρησαν στα μέλη της Επιτροπής μας χτες. Τα νούμερα αυτά πρέπει να ε, επιβεβαιωθούν σε επίπεδο Κορεπέρ και Συμβουλίου, αλλά μπορεί να κατά πάσα πιθανότητα είναι πολύ κοντά στη, στα τελικά ε, νούμερα που θα δώσει το Συμβούλιο και που, στη θέση που θα εγκρίνει στο τέλος Ιουλίου. Θέλω να κάνω λοιπόν και κάποιες επιπλέον τροπολογίες με βάση αυτά τα στοιχεία. Συνολικά η Ευρωπαϊκή Επιτροπή στο σχέδιο προπολογισμού του Απριλίου έκανε μια ρεαλιστική και επαρκή εκτίμηση των πιστώσεων που θα χρειαστούν για να καλυφθούν τα νέα αλλά και τα υφιστάμενα έργα και τα προγράμματα που θα χρηματοδοτηθούν στον τομέα της ανάπτυξης και της ανθρωπιστικής βοήθειας. Εκεί που πρότεινε περιορισμό το, της χρηματοδότησης στην ανάπτυξη, κυρίως σε είναι σε σχέση με τον DCI. Πρέπει να διατηρήσουμε τα τις πιστώσεις του 2012 σε επίπεδο δαπανών προσωπικού και για τις εξωτερικές σχέσεις και για την ευρωπαϊκή βοήθεια, το EuroPaid. Αλλιώς πώς θα, θα εξασφαλίσουμε την σωστή αξιολόγηση και τα πρότυπα. Πώς θα τα μετρήσουμε, πώς θα τη μετρήσουμε αυτή την επιτυχία. Έχω επανειλημμένως αναφερθεί στο ότι ενησυχώ για την ανάπτυξη του, των 51 ατόμων από το DCI στο DPI και αυτή η μετακίνηση της χρηματοδότησης, η ανακατανομή της χρηματοδότησης από το DCI στο EMPI. Στο Ιράν, Ιράκ και την Ιεμένη και όλα αυτά τα έχω βάλει στις προτάσεις μου. Για, την... για το περιβάλλον και την βιώσιμη διαχείριση των φυσικών πόρων και οι, τα, οι για το κλίμα και την βιοπικιλότητα είναι ασαφείς. Για να μην φύγουν οι αναπτυξιακές ε, τα αναπτυξιακά κονδύλια από ε, το χώρο της ανάπτυξης θα πρέπει να έχουμε κάτι παραπάνω από τα 46 εκατομμύρια που προτείνει η Κομισιόν. Μάλλον στα 63 εκατομμύρια ε, θα ήμασταν πιο ρεαλιστές για να εξασφαλίσουμε, να διασφαλίσουμε την προσθετικότητα της χρηματοδότησης. Δηλαδή προτείνουν τα 2-3 από ό,τι μοιάζει ότι είναι απαραίτητο. Όσον αφορά την ε, ανάπτυξη, ανθρώπινη και κοινωνική ανάπτυξη, από 40 στα 50 εκατομμύρια γίνεται πρόταση. Ένα μέρος των πιστώσεων θα χρησιμοποιηθούν για την πρόσβαση σε ε, συστήματα κοινωνικής προστασίας σε αναπτυσσόμενες χώρες. Αυτό είναι ε, χρήσιμο γιατί στο DCI προβλέπουμε ένα νέο κεφάλαιο που προσπαθεί να προσφέρει περισσότερη οικονομική ασφάλεια στους λαούς των αναπτυσσομένων χωρών. Επίσης, προτείνουμε στις τροπολογίες και ε, πιστώσεις για δημιουργία θέσεων εργασίας. Τώρα, στο σχέδιο προπολογισμού, με βάση τα προσωρινά νούμερα που κυκλοφόρησε την προηγούμενη εβδομάδα, μοιάζει ότι το Συμβούλιο περικόπτει τις προτάσεις της Επιτροπής εκ περαιτέρω. Στο DCI, οι συγκεκριμένες γραμμές προϋπολογισμού, επιστημική ασφάλεια μείων 6 εκατομμύρια σε δεσμεύσεις και μείον 4 σε πληρωμέ. μείον 38 εκατομμύρια σε πληρωμέ. μείον 15 εκατομμύρια σε πληρωμέ. παιδεία, μείον 5 εκατομμύρια σε ε, υποχρεώσεις, μείον non-state actors, μείον 5 εκατομμύρια σε υποχρεώσεις, η στήριξη για τις χώρες του πρωτοκόλου σάχαρης μείων 9 εκατομμύρια σε πληρωμές, Συνδευτικά μέτρα μπανάνες μείων 20 εκατομμύρια, ανθρωπιστική βοήθεια μείων 2 εκατομμύρια σε υποχρεώσεις, μείων 37 σε ε, πληρωμές. Αυτά κάνει δύσκολο την, στην Επιτροπή να επιτύχει τους στόχους του πολιτούς προγράμματος ε, ε, μέχρι το 2013 στους θεματικούς αυτούς χώρους και αυτό συνεπάγεται ότι θα μειωθούν πολλά πράγματα στον τομέα της υγείας, της ε, παιδείας και της αντικαταπολέμησης της πείνας τώρα στα γεωγραφικά. Η βοήθεια της Παλαιστίνης μειών 53 εκατομμύρια σε πληρωμές θα σημαίνει ότι συνολικά θα μπορέσουμε να καλύψουμε τις δαπάνες το 2013 που ήδη έχει, αν το εγκρίνει το Συμβούλιο το Αφγανιστάν, μείον 8,5 εκατομμύρια και αυτό θα στείλει αρνητικό πολιτικό μήνυμα τη στιγμή που ξεκίνησε πριν από τρεις μέρες η διάσκεψη του Τόκιο και θα δοθούν από την Αμερική εκατομμύρια δολάρια, 16 εκατομμύρια δολάρια για την ασφάλι, εξασφάλιση όταν έχουν συμφωνήσει και οι αφγανικές αρχές για νέους όρους αντιμετώπισης της ενδημικής Με την Αμερική μείον 13 εκατομμύρια 5 εκατομμύρια συνεργασία με την Κεντρική Αφρική. Αυτές οι μειώσεις πληρωμών θα επηρεάσουν τις προσπάσεις της Επιτροπής να τηρήσει τις συμβατικές υποχρεώσεις που έχει διαναλάβει. Και υπάρχει ένα, ένας, ήδη, ένας κύκλος που έχει ήδη ξεκινήσει θα πρέπει να πληρωθούν τότε και τόκοι σε καθυστερημένες, σε πληρωμές. Και το 2014, αν προτεθούν οι προτινόμενες πληρωμές περαιτέρω, αναβληθούν περαιτέρω, θα πρέπει αυτό να γίνει σε βάρος προγραμμάτων και έργων που έχουν σχεδιαστεί για το επόμενο πολιτές πρόγραμμα. Επιπλέον, οι προτάσεις του Συμβουλίου να μειωθούν τα επίπεδα πληρωμών της κατεπίγουσας βοήθειας κατά 10 δηλαδή θα πάνε στο 0. Αυτό το αποθεματικό έχει σχεδιαστεί για να μπορέσει η Ευρωπαϊκή Ένωση να ανταποκρίνεται ταχαίως σε ανθρωπιστικές ανάγκες εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης, οι οποίες όμως ήταν απρόβλεπτες στην εποχή που συντάχθηκε ο προπολογισμό. Τα τελευταία χρόνια το απόθεμα αυτό έχει χρησιμοποιηθεί για να αντιμετωπιστοποιηθούν επιπλέον ανάγκες που προέκυψαν κατά τη διάρκεια του οικονομικού έτους στο τέλος κάθε χρόνου είχε πλήρως χρησιμοποιηθεί. Έτσι, αν δεν υπάρχουν πληρωμές όταν θα υπάρξει κάποια ανθρωπιστική καταστροφή κάποιων διαστάσεων, θα επηρεάσει αυτό πολύ την ταχύτητα της αντίδρασής μας. Παράδειγμα, πρόσφατα εγκρίναμε την χρήση του για 25 εκατομμύρια για να αποκριθούμε στην επισητιστική κρίση της περιοχής του Σαχέλ. Τέλος, κυρία Πρόεδρε, αν ε, το Συμβούλιο δεν συμφωνήσει στην μετακίνηση του προσωπικού από τον DCI και στην έδρα και στις ευρωπαϊκές ε, αντιπροσωπείες θα έχουμε περαιτέρω μείωση. Αυτό σημαίνει ότι θα αυξηθεί ο χρόνος δουλειάς, ο όγκος δουλειάς. Το Κοινοβούλιο πρέπει να απαλλάσσει κάθε χρόνο την Κομισιόν για τη διαχείριση του προηγουμένου έτους. Αλλά η, μείωση, η περαιτέρω μείωση του, του προσωπικού του DCI θα επηρεάσει έτσι περαιτέρω την χρηματοοικονομική διαχείριση του DCI και κινδυνεύουμε να ξεπεράσουμε ένα όριο. Οπότε η ποιότητα αυτής της διαχείρισης να μην είναι πλέον εγγυημένη και άρα να τεθεί σε κίνδυνο η απαλλαγή δεύτερη ομάδα τροπολογιών που σύντομα θα σας στείλω ε, θα αφορά την αντιμετώπιση αυτών των περικοπών. Θα ήθελα τώρα να ακούσω τα, σχόλια των συναδέρφων για τις τροπολογίες αυτές και να υπενθυμίσω στην Επιτροπή ότι η προθεσμία υπολογής, υποβολής τροπολογιών είναι 17 Ιουλίου 5 το απόγευμα και ότι η τελική ψηφοφορία στην Επιτροπή θα γίνει στις 12 Σεπτεμβρίου. Ευχαριστώ. Ευχαριστούμε για όλα και ό,τι κάνατε για αυτό το θέμα του προπολογισμού. Ε, προοπτικές είναι λίγο ανησυχητικές σε σχέση με τα στοιχεία που μας δίνετε. Θα δώσω το λόγο στην Επιτροπή για να εκφραστεί. Όχι, όχι, όχι, κάποιος. Η κυρία θα ζητάει πρώτο λόγο. Κοιτάξτε, πριν να πάρει το λόγο η Επιτροπή, να επιμείνω σε κάτι. Εμείς σαν σοσιαλιστές δημοκράτες έχουμε την πρόθεση να καταθέσουμε κάποιες απολογίες πριν από τις 17 Ιουλίου. Θα τις έχετε σε μερικές μέρες. Θα ήθελα να σας πω ότι συμμεριζόμαστε τις εξηγήσει που έκανε ο κύριος Μίτσελ και θα ήθελα να σας πω ότι και εμείς θεωρούμε ότι βλέπουμε κάποια προβλήματα σε σχέση με τον προπολογισμό διαρθρωτικά, πράγματα τα οποία έχουμε καταγγείλει επανειλημμένως. Ορισμένα ταμεία δεν έχουν τους κατάλληλους πόρους, Αποθεματικά επίση υπάρχουν τα θέματα που έχουν να κάνουν με τι ανθρωπιστικέ κρίσει, όπω είπε και ο συνάδελφό μα, ε, κρίσεις οι οποίε είναι απρόβλεπτες, ορισμού. Δεν έχουμε κατάλληλο προπολογισμό για να αντιμετωπίσουμε κάτι τέτοιο. Και αυτό επαναλαμβάνεται. Το έχουμε επαναλημμένα θίξει, χωρί όμω να έχουμε ικανοποιητικέ απαντήσει. Οι δεσμεύσει είναι σε επίπεδο ανησυχητικό, το ίδιο και οι πιστώσει πληρωμών. Έχουμε ένα προπολογισμό που δεν ξεπερνάει, που είναι υπολείπεται σχέση με τον του 2012. Δεν είναι αποδεκτός κάτι, αυτός ο προπολογισμό. Οι παρεμβάσεις των χωρών μελών ήταν τέτοιες που μειώνανε τον προπολογισμό. Επίσης στοιχεία έχουν διαστρεβληθεί, συγκεκριμένα από τη δική μας κυβέρνηση. Αν θέλουμε δηλαδή να διατηρήσουμε την αξιοπιστία μας σε παγκόσμιο επίπεδο, θα πρέπει να προβλέψουμε πιστώσεις ε, απαραίτητες και κανές. Όταν έχουμε τέτοιο επίπεδο ε, πιστώσεων πληρωμών, δεν μπορούμε να κάνουμε σεβαστές τις δεσμεύσεις μας. Πραγματικά φέτος το επίπεδο είναι δραματικό. Ήδη υπάρχει μείωση όσον αφορά τις δεσμεύσεις, επιπλέον δεν μπορούμε να τις κάνουμε σεβαστές, καταλαβαίνετε. Το επίπεδο πιστώσεων πληρωμών είναι πολύ χαμηλό. Γι' αυτό και αντιμετωπίζουμε σε μείζωνα προβλήματα. Αυτά όσον αφορά τον προπολογισμό και πώ λειτουργεί. Τώρα, στη συνέχεια, κάποιε παρατηρήσει θα τι κάνουμε όταν φτάσουμε με τι τροπολογίε μα, όταν φτάσουμε στο θέμα του περιεχομένου. Πρόεδρο, τώρα θα δώσουμε το λόγο στην Επιτροπή. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Έχετε απόλυτο δίκιο. Ο προπολογισμός του 2013 συντάχθηκε με βάση τη λογοδοσία, τη διαφάνεια και με γνώμονα να ασφαλίσουμε ότι τουλάχιστον ευθυγραμμιζόμασταν με τον προϋπολογισμό του 2012, αν και να, αυξήσουμε λίγο σε κάποιες ε, γραμμές του προϋπολογισμού τα κονδύλια. Δεδομένου ότι ε, τηρήθηκαν οι προϋποθέσεις του πολιετούς δημοσιονομικού πλαισίου 2007-2013 παρόλο που γίνανε κάποιες προσαρμογές. Τώρα, προσπαθήσαμε επίσης να διασφαλίσουμε ότι αυτό που ζητάει η Κομισιόν σε καιρούς λιτότητας είναι το ελάχιστο απαραίτητο για να υπάρχει μια συνέχεια στην πολιτική μας, για να υπάρχει μια συνέχεια στη δουλειά μας και να μπορούμε να τηρήσουμε τις νομικές δεσμεύσεις. Βλέπουμε τώρα ότι το Συμβούλιο έχει προβεί σε περικοπές. Δεν είναι πρωτοφανές αυτό. Και στρεφόμαστε προς το Κοινοβούλιο για να εξασφαλίσουμε ότι θα δοθεί η απαραίτητη σημασία στο, στην αναπτυξιακή βοήθεια, στο εργαλείο για την αναπτυξιακή συνεργασία. Όλοι συμφωνούμε ότι πρέπει να δουλέψουμε για την επίτευξη των στόχων ε, της χιλιετηρίδας το συντομότερο δυνατό και όλοι συμφωνούμε ότι πρέπει να δουλέψουμε έτσι ώστε οι πιο μειονεκτικές πληθυσμιακές ομάδες σε όλο τον κόσμο ε, δεν τεθούν σε ακόμα μειονεκτική θέση λόγω της δικής μας οικονομικής κρίσης. Και αυτό προσπαθεί να κάνει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Βέβαια, το Συμβούλιο έχει άλλη ατζέντα ενίοτε. Δεν θέλω να υπησέλθω στο θέμα αυτό με περισσότερες λεπτομέρειες. Θέλω να σας πω ότι χαίρομαι ιδιαίτερος και με ενθαρρύνει κιόλας η πρόταση του εισηγητή και η ανάλυση την οποία κάνει δείχνοντας ότι θα πρέπει να αποκατασταθούν όλα αυτά τα οποία ήταν στα αιτήματα της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Είχαμε πολύ μεγάλα περιθώρια. Ε, πέρυσι το περιθώριο ήταν 200 εκατομμύρια ευρώ για τον προπολογισμό για την εξωτερική δράση της Ευρωπαϊκής Ένωσης και φέτος το σχέδιο προπολογισμού φτάσαμε στα 500 και με τις περικοπές στο Συμβούλιο αυξάνεται το περιθώριο τελικά. Και τελικά έχει το Κοινοβούλιο μεγαλύτερο περιθώριο ελιγμών προτού ε, θέσει τις προτεραιότητες του επιτάπητο στο Συμβούλιο, τις οποίες προτεραιότητες βεβαίως θα παρακολουθήσει προσεκτικά η Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Ελπίσουμε να έχουμε την ευκαιρία να προβάλλουμε τα ίδια επιχειρήματα και στην Επιτροπή Προϋπολογισμών του Κοινοβουλίου. Ευχαριστώ πολύ. Μάλιστα, ευχαριστούμε. Ο κύριος Μίτσελ να κλείσει. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Συμφωνώ με τα σχόλια της συναδέλφου κυρία Στόγια εκτιμώ ιδιαίτερο τι ανησυχίες τις οποίες μοιράστηκε μαζί μας. Τις καταλαβαίνω πράγματι και χαίρομαι διότι ακούω ότι το Κοινοβούλιο με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή ε, τάσσονται από την ίδια πλευρά. Η Επιτροπή ελπίζει ε, το Κοινοβούλιο να προσφέρει ισχυρή στήριξη σε αυτήν και ας ελπίσουμε ότι και τα κράτη-μέλη θα ε, το πράξουν και ότι οι μη κυβερνητικέ οργανώσει θα έρθουν σε επαφή όχι μόνο με μέλη του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, αλλά και με μέλη των Εθνικών Κοινοβουλίων. Είναι μια τριμερή προσέγγιση αυτή. Ξέρουμε ότι σε πολλά κράτη-μέλη ε, υπάρχει μια περιχαράκωση γενικότερη, αλλά αυτή η συνεισφορά το 0,7 για το GNI ε, δεν θα πρέπει να μειωθεί έτσι περαιτέρω. Πρέπει να αγωνιστούμε και είναι καλό το ότι διαπιστώνουμε ότι είμαστε ενωμένοι στη δική μας Επιτροπή και είμαστε και ενωμένοι με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Ε, ε, βέβαια, μένει πολλή δουλειά να γίνει σε επίπεδο Συμβουλίου. Θα ε, δουλέψω πάνω στις υπόλοιπε τροπολογίες και θα τις υποβάλω στην Επιτροπή. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ, λέει Πρόεδρος. Η προθεσμία κατάθεσης τροπολογιών 17 Ιουλίου στις 10 το πρωί. Περνούμε τώρα στην ενδιάμεση έκθεση με σκοπό τη θετική έκβαση της διαδικασίας έγκρισης του πολιετούς δημοσιονομικού πλαισίου. Είναι λοιπόν ένας εξαιρετικά σημαντικός φάκελος ε, για την ε, συνεργασία για αναπτυξιακά θέματα στο μέλλον και στο πλαίσιο του πολιετούς δημοσιονομικού πλαισίου 2014-2020 είναι ένα θέμα που μας απασχολεί ιδιαιτέρως. Δεδομένου ότι ε, το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο τον Οκτώβριο θα εθετήσει την επίσημη θέση του Συμβουλίου, η Επιτροπή Προπολογισμών που είναι αρμόδια επί της ουσίας για τα θέματα αυτά, αποφάσισε ε, στις αρχές Οκτωβρίου να ψηφίσει ε, την έκθεσή της, άρα νωρίτερα από ό,τι προβλεπόταν και καλούμαστε λοιπόν και εμείς νωρίτερα από ό,τι προβλεπόταν να έχουμε ετοιμάσει την γνωμοδότησή μας. Πρόκειται λοιπόν για ε, μια αρκετά ασφικτική προθεσμία για την κατάθεση των τροπολογιών σας. Κύριε Γκέρενς, ε, θα μοιραστείτε μαζί μας τις σκέψεις σας και τους προβληματισμούς σας. Να σας εφιστήσω καταρχάς την προσοχή στο γεγονός ότι ε, δεν έχουμε γραπτές μεταφράσεις ε, σε όλες τις γλώσσες ακόμα, διότι έχει μειωθεί το κονδύλιο για μεταφράσεις κατά τη διάρκεια των θερινών διακοπών και ε, ζητώ την επίοικιά σας. Κύριε Γκέρες, έχετε το λόγο. Μπορείτε να μας κάνετε την ανάλυση σας, παρακαλώ. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Το σχέδιο έκθεσης Επιτροπής προϋπολογισμών δεν είναι ακόμα διαθέσιμο. Επομένως, η γνωμοδότηση αυτή η δική μας βασίζεται στα δύο έγγραφα ε, κλειδιά της Επιτροπής σε σχέση με το επόμενο βασικό πολιετές δημοσιονομικό σχέδιο. Πρόταση κανονισμού του Συμβουλίου που προσδιορίζει το πολιετές δημοσιονομικό πλαίσιο 2014-2020 και σχέδιο ε, διαθεσμικής οργανικής διοργανικής συμφωνίας μεταξύ Κοινοβουλίου, Επιτροπής και Συμβουλίου ε, για θέματα συνεργασίας ως προς τον προπολογισμό και για τη χρηστή οικονομική διαχείριση. Θα ήθελα να σας επισημάνω ότι στις 6 ε, του Ιουλίου η Επιτροπή οθέτησε ε, μία τροποποιημένη ε, πρόταση για αυτό τον κανονισμό όπου λαμβάνεται υπόψη η συνεισφορά της Κροατίας άπαξ και προσχωρήσει η χώρα αυτή στην Ευρωπαϊκή Ένωση και όπου λαμβάνονται υπόψη και τα νέα στοιχεία ως προς το ακαθάριστο εχώριο προϊόν ορισμένων κρατών μελών διότι έχουν επανυπολογιστεί ε, όλα αυτά τα στοιχεία στο πλαίσιο της πολιτικής συνοχής και έχουν γίνει οι απαραίτητες αναγωγές στο συλλογικό ΑΕΠ της Ένωσης. Όλες αυτές οι τεχνικές προσαρμογές δεν επηρεάζουν τη χρηματοδότηση της γραμμής του προϋπολισμού υπαριθμών 4 που μας αφορά από τη στιγμή που αρχική πρόταση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής εκεί λάμβανε υπόψη της ότι μετά την προσχώρηση στην Ευρωπαϊκή Ένωση η Κροατία δεν θα είναι δικαιούχος βοήθειας βάσει της γραμμής ε, γιατί αυτή αφορά μόνο τις τρίτες χώρες. Πάμε τώρα ε, στα γενικά ε, συμπεράσματα στο περιεχόμενο αυτού του σχεδίου γνωμοδότησης. Υπενθυμίζει λοιπόν ο εισηγητής ότι η ημερομηνία κλειδί για το 2015 ε, είναι η ημερομηνία για την επίτευξη των στόχων της χιλιετηρίδας και για την επίτευξη όσων είχαν αποφασιστεί ήδη από το 2007 και το 2015 είναι το μισό της περίοδου. Αν αποσυρθούν λοιπόν κονδύλια, αυτό θα είναι αντιπαραγωγικό. Θα πρέπει η Ευρωπαϊκή Ένωση να αξιοποιήσει το επόμενο πολιετές δημοσιονομικό πλαίσιο για να προωθήσει ακόμα περισσότερο την τήρηση των διεθνών της δεσμεύσεων. Και το κύριο, το βασικό επιχείρημα για τη διατήρηση του προπολογισμού σε επαρκή επίπεδα είναι ακριβώς η ποιότητα της βοήθειας που προσφέρουμε. Πάρα πολλέ αναλύσεις έχουν γίνει. Μιλώ για την ε, έρευνα και την έκθεση του ΟΑΣΑ το 2012. Ε, μιλώ για διάφορα άλλα ερευνητικά κέντρα, τα οποία δείχνουν ότι εμείς είμαστε στην πρώτη θέση παγκοσμίω ως προς την αναπτυξιακή βοήθεια με διαφάνεια και με απτά αποτελέσματα, τα οποία τελικά ε, βελτιώνουν την ποιότητα ζωής των ε, πολιτών, των ανθρώπων που διαβιούν στις αναπτυσσόμενες χώρες. Αυτά λοιπόν είναι προς τιμήν της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Θα ήθελα να υπογραμμίσω ότι συμφωνούμε με την πρόταση της Επιτροπής για την ε, γραμμή 4, και μιλούμε για ένα εργαλείο χρηματοδότησης ε, της αναπτυξιακής βοήθειας και δεν θέλουμε όλα αυτά να θυσιαστούν ε, ε, στο βωμό της λιτότητας που επικρατεί στα κράτη-μέλη αυτή τη στιγμή. Η αρχή της διαφοροποίησης δεν μπορεί να χρησιμοποιηθεί ως πρόσχημα, ως δικαιολογία για να μειωθεί η αναπτυξιακή βοήθεια που προσφέρουμε. Η διαφοροποίηση αυτή πρέπει να οδηγεί στη συγκέντρωση της βοήθειας σε λιγότερο αριθμό κρατών που θα είναι επιλέξιμα κράτη και να μην πλήξει συνολικά ε, το DCI, το εργαλείο δηλαδή για την αναπτυξιακή συνεργασία. Θα πρέπει να έχουμε ευελιξία στη χρηματοδότηση της ε, ανθρωπιστικής βοήθειας και της αναπτυξιακής βοήθειας. Και αν το ε, αποθεματικό για επίγοντα, το οποίο είναι εκτός του γενικού προϋπολογισμού της Ένωσης, μπει τελικά στο πυρήνα του προϋπολογισμού της Ένωσης, θα τεθεί ένα αμφιβόλο αυτή η ευελιξία που έχουμε. Το αποθεματικό, το απόθεμα που έχουμε λειτουργεί πολύ καλά αυτή τη στιγμή. Δεν υπάρχει κανένας λόγος να μπει μέσα στο όριο του CFP εάν τελικά ο σκοπός δεν είναι να μειωθούν ε, οι κατανομές ε, βάσει της ε, γραμμής του προπολογισμού υπαριθμών 4 για την εξωτερική δράση της Ένωσης. Υπενθυμίζω λοιπόν ότι είναι σαφής η θέση της Επιτροπής μας για την προσθετικότητα της χρηματοδότησης ε, για τις ε, κλιματικές μεταβολές, για την επίτευξη του στόχου του 7% ανέκαθεν εμείς λέγαμε ότι οι δεσμεύσεις σε αυτό το θέμα πρέπει να είναι μια επιπρόσθετη συμφωνία μια επιπρόσθετη συνεισφορά στις δεσμεύσεις ε, που έχουν ανεληφθεί στο πλαίσιο της αναπτυξιακής βοήθειας. Και μιλώ και για την ένταξη στο προϋπολογισμό του Ευρωπαϊκού Ταμείου για την Ανάπτυξη. Δεν μπορεί να χρησιμοποιηθεί αυτό ως ε, πρόσχημα τελικά για να μειωθούν οι δυνατότητες. Αυτό το επιθυμούν ορισμένοι κράτη-μέλη. Και θα έλεγα ότι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή πρέπει να υποβάλει προτάσεις για την ενίσχυση του δικαιώματος ελέγχου του Κοινοβουλίου σε, όλες αυτές, σε όλο αυτό το πλαίσιο συνεργασίας με τις ε, χώρες ΑΚΕ. Κάτι το οποίο έχει γίνει επανειλημμένος. Και τέλος, ε, θα ήταν ενδιαφέρουσα και η άποψη του Συμβουλίου για αυτό το ε, θέμα. Καλείται η Ευρωπαϊκή Επιτροπή να ε, περιλάβει αυτά στον κεντρικό προϋπολογισμό στο επόμενο πολιετές δημοσιονομικό πλαίσιο, όχι μόνο σε αυτό 2014 με 2020, αλλά και στο 2020 και μετά τελικά στις 3 Σεπτεμβρίου μπορούμε να ε, ψηφίσουμε στην Επιτροπή μας την ε, έκθεση αυτή. Και σας ευχαριστώ πολύ για την ε, αμέριστη προσοχή σας, η Πρόεδρος. Ευχαριστώ, ο κύριος Κορτές Λάστρα. Ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε. Θέλω να ευχαριστήσω τον Σάγλε για την πολύ καλή δουλειά του κατάφερε να συμπεριλάβει τα θέματα που μας απασχολούν περισσότερο από όλα εν ώψη του επόμενου πολιετούς δημοσιονομικού πλαισίου 2014-2020. Χρειαζόμαστε ένα τέτοιο πλαίσιο να είναι πολύ φιλόδοξο. Εκατομμύρια παιδιά δεν μπόρεσαν να πάνε σχολείο. Ε, νομίζω όμως ότι η δική μας δουλειά έχει ε, πάρα πολύ μεγάλα ωφέλη γιατί 5 ε, εκατομμύρια παιδιά εμβολιάστηκαν, δεκάδες άλλα απέκτησαν πρόσβαση σε σωστές συνθήκες ίδρυυσης και υγιεινής και πολλά εκατομμύρια άλλα παιδιά τελικά μπόρεσαν να πάνε σχολείο. Αυτά, όλα αυτά δείχνουν τα αποτελέσματα της δουλειάς μας. Χρειαζόμαστε λοιπόν μεγαλύτερο συντονισμό για να είναι πιο αποτελεσματική η βοήθειά μας και ε, αυτό θα μπορούσε να βοηθήσει τα κράτη μέχρι και το ποσό των 5 εκατομμυρίων ευρώ ετησίως. Και πρέπει να καλύψουμε και το κενό των 47 εκατομμυρίων ευρώ που μας λείπει για να πετύχουμε το στόχο του 0,7%. Ο εισηγητής ε, μας παρουσίασε ε, εξαιρετικά το όραμα της Επιτροπής. Δεν μπορούμε να δεχθούμε τις περικοπές. Τα αποτελέσματα και η προστιθέμενη αξία της αναπτυξιακής βοήθειας είναι πράγματα πασιφανή, αποδεδειγμένα και θα πρέπει να δοθούν τα μέσα για να επιτύχουμε τις προσδοκίες μας. Δεν θα δεχθούμε περικοπές στο εργαλείο, στο μέσο για την αναπτυξιακή συνεργασία. Ναι, πρέπει να συγκεντρώσουμε τους πόρους μας και σταδιακά να βγουν από αυτό το εργαλείο οι χώρες που πληρούν τις δεσμεύσεις του Μπουσάν ε, και τις εταιρικές σχέσεις, δηλαδή του Πουσάν. Και θα ήθελα να πω ότι θα υποβάλω τροπολογίε σε σχέση με την επιβολή φόρου χρηματιστηριακών συναλλαγών, ο οποίο θα μπορούσε να οδηγήσει ε, τα χρήματα αυτά να χρησιμοποιηθούν για την αναπτυξιακή βοήθεια. Ευχαριστώ πολύ. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θα πάρει τώρα το λόγο. Παρακαλώ. Ευχαριστώ. Ε, η Επιτροπή ευχαριστεί τον κύριο Γκέρενς για τη γνωμοδότησή του. Συμμεριζόμαστε σε γενικές γραμμές ότι έχει διαπιστώσει να μην χρονοτριβήσω όμως δημιουργούνται κάποιοι προβληματισμοί σε σχέση με αυτές τις διαπιστώσεις. Έχουμε το δικαίωμα φυσικά εδώ πέρα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και η Κομισιόν επανειλημμένα έχει κάνει επανειλημμένα δείξει τη διάθεσή της να βελτιωθούν οι, οι συνεργασίες μας. Αυτό το η δυνατότητα δηλαδή να μπορεί να έχει μια άποψη το Κοινοβούλιο γίνεται σεβαστή από την Κομισιόν. Θεωρούμε ότι μπορεί να γίνει ένας διάλογος άτυπος ούτω ώστε να βελτιώσουμε τη συνεργασία μας για τον προπολογισμό που θα κρυφθεί για το 2013. Θα ήθελα να ξαναευχαριστήσω τη συμβολή του Κοινοβουλίου όσον αφορά τώρα ότι για το θέμα που έχει να κάνει με τη θέση της Επιτροπής εμείς αυτό που θέλουμε να πούμε ότι έχουν γίνει πολύ λεπτές διαπραγματεύσεις σε πλαίσια της συμφωνίας για το Κοτονού νομικά είναι πολύ δύσκολο να κάνει κάποιες κάποια αλλαγή σε αυτά τα πλαίσια των διαπραγματεύσεων. Εμείς όμως θα επανέλθουμε για την περίοδο 2014-2020 διότι η Επιτροπή θα αναλάβει να προβληματιστεί γενικά σε σχέση με την δομή που έχει να κάνει με τη συνεργασία της Ευρωπαϊκής Ένωσης και της χώρας ΑΚΕ και θα κοιτάξει να κάνει συγκεκριμένες προτάσεις όσον αφορά τον προϋπολογισμό. Τώρα για το DCI, κλείνοντα κλείνοντας, θα πω ότι συμμεριζόμαστε τις διαπιστώσεις του κυρίου Γκέρενς εμείς επανειλημμένα έχουμε εκφραστεί σε αυτό το θέμα σε σχέση για τις προβλέψεις που έχουν γίνει. Δεν υπάρχει κανένα πρόβλημα. Να μην πω τώρα στις λεπτομέρειες. Είναι αρμοδιότητα που έχει να κάνει με τις χώρες μέλη. Να δούμε τώρα στα πλαίσια τώρα και της γενικότερης κρίσης αν μπορεί να υπάρξει κάποια λύση όλοι και οποιασδήποτε αλλαγέ μπορέσουν να γίνουν είναι, μπορούν να τις δούμε με μια σχετική επιφύλαξη. Ευχαριστώ. Πρόεδρος, σας ευχαριστώ πολύ. Ο κύριος Γκέρος μήπως θέλει να κλείσει τώρα, να πάρει πάλι το λόγο να κλείσει το θέμα. Ευχαριστώ. Μερικές παρατηρήσεις πριν να κάνω τα σχόλια. Να ευχαριστήσω τους ε, προλαλήσαντες για την έκθεσή μου Πρώτο. Για την ομοδότηση, Για την ε, τίτλο 4. Σε σχέση με την ανάπτυξη. Η Επιτροπή μου είπε σαν μια πρώτη αντίδραση στο σχέδιο που είχα καταθέσει ότι δεν ήμουν αρκετά απαιτητικό. Και πραγματικά τότε αποφάσισα να μην ξαναεκτεθώ σε τέτοια, σε τέτοιες, σε τέτοια σχόλια. Λοιπόν, θέλησα να είμαι πιο απαιτητικός. Δεν μου, το κάνει, δεν μου κάνει κάποια τέτοια παρατήρηση η Επιτροπή, άρα είμαι στη σωστή κατεύθυνση. Δεύτερη παρατήρηση. Την ε, προσθετικότητα. Αυτό που λέτε ε, ε, δεν πάει προς τη σωστή κατεύθυνση. Βλέπουμε τις χώρες μέλη που έχουν κάποιες επιφυλάξεις όσον αφορά τη βοήθεια για την ανάπτυξη. Το βλέπουμε και τα στοιχεία που παρουσιάζονται εδώ Βλέπω εδώ κάποιες διορθώσεις προς τα πάνω, αλλά απ' την άλλη έχουν γίνει κάποιες μειώσεις. Αν έχω καταλάβει, βλέπουμε εδώ πέρα πολύ συγκεκριμένα δύο-τρεις μειώσεις, αν δεν κάνω λάθος. Μια τρίτη παρατήρηση για την ΦΕΔ και τον προπολογισμό αυτής. Έχουν γίνει κάποιες προτάσεις, το λαμβάνουμε υπόψη, σίγουρα, αλλά για τη Fed, όπως είπα και πριν από λίγο, είναι κάτι το οποίο δεν έχει επαληθευτεί, γίνονται ανακοινώσει χωρίς να υπάρχει μια κάτι στην πράξη. Εγώ θεωρώ ότι είναι κάποιο θετικό στοιχείο, τουλάχιστον ότι έχουμε μια δήλωση. Τα, το Αναπτυσιακό Ταμείο της Ευρωπαϊκής Ένωσης θα ε, περάσει σε επίπεδο προπολογισμού είναι θετικό και θα το δούμε, στη, θα μπει στην, θα λέγαμε στην πραγματικότητα των χωρών ΑΚΕ. Ε, και αν αυτό γίνει στη συνέχεια, προς το 2020 και μετά θα είναι ένα θετικό βήμα σε σχέση με τις σχέσεις που έχουμε με τις χώρες ΑΚΕ Ευρωπαϊκή Ένωση. Θα ήθελα να πω δηλαδή ότι μπορεί να δει κανεί μια θετική ανάγνωση του όλου κειμένου. Και το μόνο που μπορώ να κάνω είναι να ευχαριστήσω για αυτό το επικοδομητικό πνεύμα. Πρόεδρος, υπενθυμίζω, κατάθεση πρωτοπολιών προθεσμία, Παρασκευή, 20 ε, Ιουλίου, στις 12. Συνεχίζουμε το 13, το 13ο θέμα της ημερήσιας διάταξης έχουμε να κάνουμε με ένα μηχανισμό για την πολιτική προστασία της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Έχουμε ένα νομοθετικό σχέδιο. Είχαμε μια πρώτη ανταλλαγή απόψεων ε, με τον κύριο Σέρενσεν για τη δημιουργία ενός νέου μηχανισμού της πολιτικής προστασίας στην Ευρωπαϊκή Ένωση η συζήτηση που έχουμε σήμερα έχει να κάνει με το σχέδιο γνωμοδότησης το οποίο ετοίμασε η κυρία Στρίφλερ. Να υπενθυμίσω ότι η δική μας η Επιτροπή σύμφωνα με το άρθρο 50 του κανονισμού συνεργάζεται με την Επιτροπή για το Περιβάλλον που είναι η αρμόδια ε, Επιτροπή ε, Εδώ έχουμε να κάνουμε θέματα που έχουν να κάνουν με την πολιτική προστασία και τα, την ανθρωπική βοήθεια Αυτά μας δίνουν τη δυνατότητα να έχουμε μια στενή συνεργασία με την φίλη ε, Επιτροπή. Θα δώσω αμέσως το λόγο στην κυρία Στρίφλερ τώρα. Ευχαριστώ κυρία Πρόεδρε, αγαπητοί συνάδελφοι, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο πάρα πολλές φορές ζήτησε από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή να, κάνει, να πάρει πρωτοβουλίες για να μπορέσει η Ευρωπαϊκή Ένωση να δράσει σε περίπτωση που έχουν, ε, έχουμε κάποια καταστροφή και να το κράξει αυτό με αποτελεσματικότητα. Ευχαριστώ την Επιτροπή που ανταποκρίθηκε στις αιτήματα του Κοινοβουλίου όταν είχαμε ανταλλαγή απόψεων νωρίτερα. Είδαμε, ζητήσαμε την Ευρωπαϊκή Επιτροπή να ενισχύσει το νομοθετικά το υπάρχον σύστημα. Έχουμε το άρθρο 50 όπου κάνουμε γνωμοδότηση, δηλαδή διαδικασία ε, με, τη, με τις άλλες επιτροπές οι οποίες είναι αρμόδιες και έχουν κοινέ ε, αρμοδιότητες αυτό το άρθρο που μας αφορά απαιτεί, ε, σημαίνει ότι πρέπει να ενισχυθεί αυτή η συνεργασία. Όταν έχουμε ε, καταστροφές λόγω ανθρωπίνης λόγου, ε, υπάρχει ένα προβληματισμό. υπάρχουν κάποιοι συγκεκριμένοι κανόνες με τις οποίες επεμβαίνει κανείς, είναι διαφορετική η πολιτική προστασία όταν είναι ο ανθρώπινος παράγοντας ή όταν είναι φυσική καταστροφή. Έχουμε ένα κεφάλαιο για το, τις δράσεις που μπορούν να γίνουν για, το, για τις προετοιμασίες που μπορούν να γίνουν. Έχουμε τη δυνατότητα να χρηματοδοτήσουμε δράσεις πρόληψης και προετοιμασίας σε χώρες που έχουν ανάγκη και σε ειδικέ περιπτώσεις, όπως στην Αιτία για παράδειγμα, ε, έχουμε μια χώρα η οποία πολύ συχνά έχει πληγεί. Εδώ έχουμε να κάνουμε την ικανότητα της Ευρωπαϊκής Ένωσης να δράσει σε επίγοντα κατάσταση και να γίνει με το σωστό τρόπο σε σχέση με την αρχή που αφορά την πολιτική προστασία, να το κάνει αυτό με, στρατιωτική, ε, με στρατιωτικό τρόπο ή με οικονομικά μέσα. Η, ε, αυτό που μετράει είναι αποτελεσματικότητα, αλλά χρειάζεται να γίνει πολλή δουλειά όσον αφορά τη διαφάνεια. Το έχουμε πει επανελειμμένα αυτό. Η Ευρωπαϊκή Ένωση θα πρέπει να έχει ή να υπαρούσα σε εθνικό και ευρωπαϊκό επίπεδο έχουμε να κάνουμε την ανθρωπική βοήθεια και την ανάπτυξη και εδώ αυτό που δεν βλέπουμε συχνά είναι δεν υπάρχει συντονισμός, χρειάζεται μια συμπληρωματικότητα. Η πολιτική προστασία μπορεί να συμβάλλει, να βοηθήσει σε δράσεις οι οποίες μπορούν να γίνουν στα πλαίσια της ανάπτυξης. Στα πλαίσια του 2014-2020 έχουμε το θέμα της συγχρονατοδότησης, στις μεταφορές, και εδώ έχουμε το άρθρο 23 σε σχέση με την απόφαση, έχουμε ενίσχυση των δράσεων πρόληψης και προετοιμασίας εν ώψη γεγονότος, δράσεις σε σχέση με το άρθρο 2021. Έχουμε να κάνουμε την πολιτική γυτνίαση σε ευρωπαϊκό επίπεδο και συμμετοχή σε μηχανισμούς αντιμετώπιση περιπτώσεων αναπερίπτωση για τη βοήθεια χωρών που βρίσκονται σε ανάγκη. Λιγότερο ανεπτυγμένες. έχουμε δράση η οποία έγινε εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης και η οποία αντιμετώπισε με άνισο τρόπο τις διάφορες περιπτώσεις. Για το 2014-2020 θα πρέπει ε, η δράση μας να αντικατοπτρίζει την πραγματικότητα που έχουμε μπροστά μας. Ευχαριστώ πολύ. Ζητήσατε το λόγο. Ναι. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Τα τελευταία χρόνια οι καταστροφές στην Αϊτή και στο Πακιστάν μας υποθύμησαν πόσο δύσκολο είναι να μπορεί να υπάρξει ευρωπαϊκός συντονισμός και να μπορέσει η δράση της ε, Ένωσης να είναι σαφής. Το άρθρο της Συνθήκης για τη Λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης μας δίνει σήμερα την ευκαιρία να ενισχύσουμε την ευρωπαϊκή δυνατότητα πρόληψης και προστασίας των φυσικών, από τις φυσικές καταστροφές ή τις ανθρωπογενείς καταστροφές στο εσωτερικό και στο εξωτερικό της Ένωσης. Η Ευρωπαϊκή δεν ε, δίνει λευκή σελίδα, αλλά προσπαθεί να εξορθολογήσει τους υφιστάμενους κανονισμούς. Πράγμα που θα ολοκληρωθεί με την ε, υιοθέτηση του κανονισμού πέρα από αυτά που γίνονται τώρα, αυτό που πρέπει να καθοδηγεί την εργασία της δουλειάς μας από αυτού είναι η συνοχή ανάμεσα σε αυτή την πρόταση και την Ευρωπαϊκή Συνένεση για την ανθρωπιστική βοήθεια. Έχουμε με ικανοποίηση σημειώσει ότι η ευρωπαϊκή δυνατότητα ανταπόκρισης στις κατεπίγουσες περιπτώσεις ε, θα πρέπει να μας επιτρέψει να περάσουμε από ένα σύστημα κατά περίπτωση σε ένα σύστημα που θα επαληθεύει ε, την κατάσταση με βάση ε, διαρκής, διαρκή ενημέρωση. Κατά την πρώτη ανταλλαγή απόψεων ε, δόθηκαν κάποιες διευκρινήσεις και έγιναν βελτιώσεις στον κανονισμό. Και θέλω να συγχαρώ τον εισηγητή για το εξαιρετικό του έργο που έλαβε υπόψη περισσότερες παρατηρήσεις μας. Η τροπολογία 3 της κυρίας Τρίφλερ υπενθυμίζει ότι αν το μέσο στρατιωτικό κόστος είναι αντίστοιχο με το κόστος της ανθρωπιστικής βοήθειας θα πρέπει να γίνεται σεβαστή η συμφωνία του Όσλο. Θα πρέπει να ξεκαθαριστεί και η ορολογία όσον αφορά τη διάφορα είδη καταστροφών, γιατί οι κανόνες παρέμβασης είναι διαφορετικοί. Η συγγήτρια έκανε αυτή τη διάκριση. Επίσης η πολιτική προστασία είναι σημαντικό στοιχείο προστασίας της, ε, στις φυσικές καταστροφές εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης και βεβαίως ε, τα πράγματα σε αυτές τις περιπτώσεις είναι πολύ πιο λεπτά. Δεν έχει γίνει διάκριση ανάμεσα στις δύο αυτές καταστάσεις. Η τροπολογία 12 που προτείνει η συγχύτρια διορθώνει την κατάσταση γιατί υπενθυμίζει το σεβασμό των ε, αρχών της ουδετερότητας κλπ. Ο, ο κανονισμός δεν είναι πολύ σαφής όσον αφορά τη σημασία της ανθρωπιστικής βοήθειας και της αναπτυξικής βοήθειας σε περιπτώσεις ε, καταστροφών σε αναπτυσσόμενες χώρες. Η συγκύκλια όμως θέτει, ε, δίνει έμφαση στη, στα θέματα του κατεπήγοντος της αποκατάστασης. Θα ήθελα να προτείνω μια τροπολογία προς την εισηγήτρια που αφορά την σημαντική βελτίωση της ικανότητας προστασίας σε περιπτώσεις καταστροφών εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης. Όπως γνωρίζουμε, η γεωστρατηγική θέση της Ένωσης είναι εξαιρετική λόγω των εξόχως ε, περιφερειακών περιοχών και έτσι θα ήθελα να προτείνω να δώσουμε ε, να προβλέψουμε στις περιοχές αυτές ε, ανθρώπινη και υλική βοήθεια. Ευχαριστώ πολύ. Το λόγο τώρα έχει η Επιτροπή, ο κύριος Χανστάς. Ευχαριστώ πολύ κυρία Πρόεδρε. Αρχικά θέλω να ευχαριστήσω την Επιτροπή και κυρίως την εισηγήτρια για την ε, υποστήριξη σε αυτό το πολύ σημαντικό νομοθέτημα. Με χαρά διαπιστώνουμε ότι η Επιτροπή συμφωνεί με τους βασικούς στόχους και τους σκοπούς του κειμένου και με τα χαρά διαπιστώνουμε ότι οι απόψεις του Κοινοβουλίου συνάδουν με τη, συμφωνούν με τις απόψεις των πολιτών. Το τροβαρόμετρο πρόσφατα έδειξε ισχυρή στήριξη από πλευράς πολιτών για μεγαλύτερη ελληνική στα κράτη-μέλη σε περίπτωση φυσικών καταστροφών αλλά και σε άλλες χώρες. Λοιπόν, υγιής αυτή η βάση και σαφώς είναι ευπρόσδεκτες οι διευκρινήσεις της εισηγήτριας. Η αύξηση του αριθμού των καταστροφών τόσο εντός όσο και εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης σαφώς απαιτούν ενίσχυση των μέσων που υπάρχουν για την αντιμετώπιση, την πρόληψη και την διαχείριση αυτών των καταστροφών. Μια-δυο διευκρινήσεις θέλω να κάνω σε αυτή τη φάση δεν θα κάνω τίποτα άλλο. Πρώτον, ο Ευρωπαϊκός Μηχανισμός Πολιτικής Προστασίας αποτελεί φυσικά πλαίσιο συνεργασίας κυρίως για την προετοιμασία ε, και την, ανταπόκριση καταστροφών εντός Ευρωπαϊκής Ένωσης, αλλά όπως σωστά επεσήμενε η συγγήτρια, χρησιμοποιείται επίσης, είναι πολύ χρήσιμος και για την αντιμετώπιση ε, καταστροφών εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης σε ε, συνέργεια με τα μέσα ανθρωπιστικής βοήθειας, όπως στην περίπτωση της Λιβύης πέρυσι. Είδαμε ότι και τα δύο μέσα είναι συμπληρωματικά και τα δύο μπορούν να ε, ε, συγχρησιμοποιηθούν για την αντιμετώπιση κατεβούσων καταστάσεων. Συμφωνούμε την Επιτροπή ότι είναι χρήσιμο να αναφερόμαστε στην ευρωπαϊκή συνένεση, συναντήληψη επ' αυτού και να υπάρχει διάκριση ανάμεσα στις φυσικές καταστροφές αφενός και τις ε, σύνθετες κατεβίουσες καταστάσεις από την άλλη. Τροπολογία παριθμών 10. Θα ήθελα να σημειώσω ότι απαιτούνται μεγάλες δαπάνες στο κεφάλαιο 3 του προϋπολογισμού για να μπορέσουμε να αποκριθούμε σε κατεπίγουσες καταστάσεις τόσο εντός όσο και εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης. Πρακτικό παράδειγμα, επενδύουμε ε, πολλά στην κατάρτιση και τις ασκήσεις εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης. Θα χρειαστούν ε, δαπάνες για την ανάπτυξη της δυνατότητας ανταπόκρισης ε, κατεπίουσες καταστάσεις ε, και πρέπει να επενδυθούν ε, πολλά σε εξοπλισμό εντός και εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης. Και γι' αυτό η Επιτροπή πρότεινε αρχικά ένα μεγαλύτερο, ελαφρώς μεγαλύτερο μερίδιο χρηματοδότησης στο κεφάλαιο 3 για αυτόν τον σκοπό εντός Ευρωπαϊκής Ένωσης. Στο σημείο αυτό θα σταματήσω. Επαναλαμβάνω όμως την ευγνωμοσύνη της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για το έργο της Επιτροπής και της εισηγήτριας σχετικά και προσβλέπουμε στη στενή μας συνεργασία στη συνέχεια αυτής της προσπάθειας. Merci Το λόγο τώρα πάρει Στρίφλερ για να κλείσει. Ευχαριστώ, ευχαριστώ για τη συμμετοχή, τα σχολιά σας. Τίποτα δεν έχω να προσθέσω. Πρόεδρος, Υπενθυμίζω, προθεσμία κατάρτισης τροπολογιών είναι η 3η Σεπτεμβρίου, το μεσημέρι, 12 η ώρα. Λοιπόν, να γίνει ίσως καλύτερα πριν την ε, πάτε για διακοπές. Λοιπόν, στο 14ο σημείο της ημερήσιας διάταξης έχουμε να κάνουμε με την έκθεση της κυρίας Σνίμπερ Γιάνστραμ έκθεση για τη συνοχή της αναπτυξιακής πολιτικής. Αποτελεί συνέχεια στη συζήτηση που είχαμε στην τελευταία συνεδρίαση, όπου η κυρία Σνίμπερ Γιάστρα μας παρουσίασε το κείμενό της. Παρακαλώ την εισηγήτρια να πάρει το λόγο και να μας παρουσιάσει τα βασικά στοιχεία του σχέδιου έκθεσης που έχει. Danke, Frau Vorsitzende, liebe Kolleginnen und Kollegen, liebe Gäste. Ich darf Αγαπητοί συνάδελφοι, αγαπητοί προσκεκλημένοι, θα ήθελα να σας παρουσιάσω την έκθεση για τη συνοχή της ευρωπαϊκής πολιτικής για την αναπτυξιακή βοήθεια. Είναι πράγματι μία από τις πιο μεγάλες προκλήσεις που πρέπει να αντιμετωπίσουμε σε θέματα αναπτυξιακής ε, πολιτικής. Ως προς το PCD θέλουμε να δούμε πώς μπορούμε να εξασφαλίσουμε την αναπτυξιακή πολιτική στο μέλλον. Το PCD είναι η πολιτική του μέλλοντος. Μόνο έτσι μπορούμε να δημιουργήσουμε πραγματικά εταιρικέ σχέσεις με τις αναπτυσσόμενες χώρες. Θα ήθελα να υπογραμμίσω ξανά ότι εμείς οι Ευρωπαίοι χρειαζόμαστε τις αφρικανικές πρώτες ύλες και όχι το αντίθετο. Εξού και έχει τόσο μεγάλη ε, σημασία το θέμα αυτό αν λάβουμε υπόψη μας και την οικονομική κρίση που αντιμετωπίζουμε. Μπορούμε λοιπόν να ε, ξεπεράσουμε αυτό το στενό ε, πλαίσιο θεώρησης που είχαμε μέχρι τώρα. Η κρίση δείχνει ότι χρησιμοποιούμε και αξιοποιούμε σωστά τις πιστώσεις που έχουμε στη διάθεσή μας. Με αυτόν τον τρόπο μπορούμε να ε, δημιουργήσουμε τις προϋποθέσεις ώστε ε, και τα κράτη και οι κυβερνήσεις ΑΚΕ να έχουν τη δυνατότητα να σημειώσουν ε, επιτυχίες. Αγαπητοί συνάδελφοι, η... Ο απολογισμός για τα δύο τελευταία χρόνια δεν ήταν καθόλου εύκολος και είναι πολύ δύσκολο όλα αυτά να ε, εκτείνονται μόνο σε τέσσερις σελίδες. Προσπάθησα να συγκεντρώσω όλα τα στοιχεία που έλαβα. Είναι πάρα πολλές οι πληροφορίες και γι' αυτό ξεπεράσαμε το, τα όρια. Όμως, άξιζε πραγματικά τον κόπο να συμπεριλάβουμε όλες αυτές τις αναφορές και γι' αυτό αποφάσισα να θέσω υπόψη σας και τις τροπολογίες για να αποφασίσετε ποια άλλα θέματα θέλετε να συμπεριληφθούν. Με αυτή τη διαδικασία ελπίζω ότι θα είμαστε σε θέση ε, να αποφύγουμε ε, τις επικαλύψεις. Το σημαντικό είναι να ξέρουμε πώς θα εδραιώσουμε το θεσμικό πλαίσιο ώστε τελικά ε, η ΣΑΠ να εφαρμοστεί στην πράξη. Η συνοχή της αναπτυξιακής πολιτικής δηλαδή. Και το βασικό επιχείρημα είναι να έχουμε πιο μακροπρόθεσμο ορίζοντα. Κατά την άποψή μου, αυτό το οποίο έχει σημασία είναι η θέση που θα υιοθετήσουμε ε, στο πλαίσιο του ε, Ταμείου για την Περιφερειακή Ανάπτυξη. Πρέπει να έχει συνοχή η πολιτική μας, περιλαμβάνοντας τις γυναίκες, την εκπαίδευση, ε, όλα αυτά είναι εξαιρετικά σημαντικά στοιχεία και γι' αυτό τα διατήρησα στο κείμενο ε, προκειμένου να τα επανεξετάσουμε και ε, στις τροπολογίες. Αναφέρομαι βεβαίως και στους στόχους τους αναπτυξιακούς μετά το 2015 και αυτό είναι εξαιρετικά σημαντικό ζήτημα για να διασφαλίσουμε τη συνοχή στην αναπτυξιακή μας πολιτική. Ήδη έχει επιτύχει πολλά η Ευρωπαϊκή Ένωση και θα πρέπει να την επενούμε γι' αυτό, αλλά θα πρέπει να επικρίνουμε και τα αδύναμα σημεία. Διότι η συνοχή της αναπτυξιακής πολιτικής είναι μία άσκηση μόνιμη αναθεώρησης και επανεξέτασης των πολιτικών μας και γι' αυτό και περιμένω τις δικές σας προτάσεις και υποδείξεις. Ευχαριστώ. Η Πρόεδρος και εγώ σας ευχαριστώ. Το λόγο έχει ο κύριος Γκέρετς. Ευχαριστώ κυρία Πρόεδρε. Θα ήθελα να ευχαριστήσω την εισηγήτρια θερμά για τη δουλειά που έκανε. Πολύ ουσιαστική, πολύ ουσιαστική δουλειά, πολύ ποιοτική δουλειά και θα αποτελέσει και το, το γνώμονα για τη δουλειά μας σήμερα αλλά και αύριο. Εξαιρετικά ενδιαφέρον στο πλαίσιο αυτή της συζήτησης είναι το εξής. Η άρνηση ε, Σύνταξη γνωμοδότησης για τη συνοχή της πολιτικής. Η Επιτροπή Εξωτερικών Υποθέσεων αποφάσισε να μην συντάξει γνωμοδότηση. Θέματα ασφάλειας, όλα αυτά τα θέματα ασφάλειας, στρατιωτικής και άλλης πρέπει να αφορούν την Επιτροπή. Ε, δεν καταλαβαίνω γιατί αρνούνται να συντάξουν γνωμοδότηση. Ε, στην Ίντα επίσης Γιατί αυτή η ε, Επιτροπή αποφάσισε με συντάξει γνωμοδότηση. Η Ήτρε το ίδιο, η Επιτροπή Γεωργία το ίδιο, η Επιτροπή Νομικών Θεμάτων το ίδιο. Όλε αυτέ οι επιτροπέ αποφάσισαν να μην συντάξουν γνωμοδότηση. Νομίζω ότι η συνοχή στις εργασίες ε, του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου θα πρέπει να ξεκινήσει από το να συνειδητοποιήσουμε όλοι μας ε, τι συνεπάγεται κάθε μία από τις δράσεις μας. Αν συνεχίσουμε κατακαιρματίζοντας και κατανέμοντας τις δραστηριότητες μόνο, δεν θα έχουμε ένα συνολικό τελικό αποτέλεσμα. Θα πρέπει λοιπόν να γίνει αυτή η διαπίσταση και να το θέσουμε υπόψη στις υπόλοιπες επιτροπές. Εδώ βεβαίως μας αφορά εξ αρχής ε, το αντικείμενο αυτό. Νομίζω όμως ότι η αρχιτεκτονική δομή της λήψης των αποφάσεων στο κοινοβούλιο μας θα πρέπει ε, να λάβει υπόψη της αυτό το στοιχείο της αλληλεξάρτησης. Αυτό κατά πρώτο λόγο. Κατά δεύτερο λόγο. Νομίζω ότι καλό θα ήταν να έχουμε σαφή στοιχεία και σαφή τοποθέτηση. Το είπα και χθες όταν σχολίασα τη μελέτη που παρουσιάστηκε για την κοινή γεωργική πολιτική. Ορισμένες μελέτες έχουν την τάση, τίνουν να επισημαίνουν στοιχεία χωρίς να τα διευκρινίζουν. Εκεί όπου μπορούμε να έχουμε ακρίβεια στα στοιχεία θα πρέπει να το απαιτούμε αυτό. Και θα ήθελα τέλος να επαναλάβω αυτό που είχα ζητήσει σε περασμένη συνεδρίαση όταν συζητήσαμε για πρώτη φορά το θέμα της συνοχής της πολιτικής ε, με την εισηγήτρια, της συνοχής της αναπτυξιακής πολιτικής, θα ήθελα λοιπόν να ξαναπώ το εξή: Στο μέλλον καλό θα ήταν να επικεντρωθούμε σε συγκεκριμένες πτυχές. Βεβαίως να γίνεται κάποιο γενικό σχόλιο, γενικές παρατηρήσεις για τη συνοχή των πολιτικών, αλλά να επικεντρώνουμε το ενδιαφέρον μας σε ορισμένα ε, θέματα για να τα προωθούμε ακόμα καλύτερα. Για παράδειγμα, για αυτή τη χρονιά θα μπορούσαμε να επιλέξουμε να επικεντρωθούμε σε ό,τι έχει σχέση με το ορίο συν 20 και ενδεχομένως να αποφασίσουμε ότι του χρόνου θα ασχοληθούμε περισσότερο με κάποιο άλλο πεδίο, κάποιο άλλο θέμα, το οποίο θα, είναι, ε, θα αφορά περισσότερο την επικαιρότητα του 2013, όπως το ορίο 20 είναι θέμα της επικαιρότητα φέτος. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ πολύ. Το λόγο έχει ο κύριος ε, Τυρολιάν. Ευχαριστώ. Ε, την εισηγήτρια για την εξαιρετική δουλειά της. Η ποιότητα της έκθεσης αποτελεί εξαιρετική βάση εργασίας. Θέλω να κάνω απλώς μερικές παρατηρήσεις. Πρώτον, όσον αφορά το θεσμικό πλαίσιο. Παράγραφος 3 είναι πολύ σημαντική υπενθυμίζεται ότι αν δεχθούμε θετικά το πρόγραμμα δράσης για την αλλαγή, αυτό θα πρέπει να επηρεάσει και άλλα σημεία του κανονιστικού πλαισίου του ήδη υπάρχοντας. Η συμφωνία, πρέπει, η συμφωνία του Κοτονού πρέπει να γίνει σεβαστή και στο πνεύμα και στο γράμμα. Σημειώνω με χαρά ότι η μόνιμη η συγγήτρια υπογραμμίζει την ανάγκη συντονισμού και διευκρίνηση των ρόλων μεταξύ του SEA e στα πλαίσια της ε, συνοχής για τις αναπτυξιακές πολιτικής. Παράγραφο 6 του σχεδίου έκθεσης επισημαίνει τον κυρίαρχο ρόλο που πρέπει να παίξει η Ένωση όσον αφορά τη συνοχή των πολιτικών για τις χώρες ΑΚΕ. Θέλω να προσθέσω πως είναι σημαντικό ο σεβασμός του άρθρου 12 της Συμφωνίας Κοτονού που ε, υποχρεώνει την Κομισιόν να ενημερώνει τη Γραμματεία των ΑΚΕ όταν κάτι γίνεται που επηρεάζει τα συμφέροντα των κρατών ΑΚΕ. Όσον αφορά το Προεδρείο της ε, Κοινοβουλευτικής Συνέλευσης ΑΚΕ Ευρωπαϊκής Ένωσης, Θυμίζω αυτά που υπο, υποθήσαμε εδώ. Θα πρέπει να υπάρχει επικοινωνία και με αυτόν τον τρόπο αυξάνει η ευαισθητοποίηση της ΑΚΕ σε σχέση με τις δυσκολίες της συνοχής. Όσον αφορά την τομεακή πολιτική επί της ουσίας για την ανάπτυξη, όπως και η συγγήτρια, λυπάμαι για την αλογιστική χρήση και την περιοριστική χρήση που κάνει η Κομισιόν του κριτηρίου ΑΕΠ κατά κεφαλή. Πρέπει να χρησιμοποιηθούν και άλλα μέτρα, άλλοι τρόποι μέτρηση του, του επίπεδου ζωής που να αντικατοπτρίζουν την πραγματικότητα χωρών ενδιάμεσου εισοδήματο για τι εμπορικέ σχέσει θα ήταν καλό να, να προσθεθεί μια παράγραφος για την ε, υπομεταρρύθμιση, αναδιατύπωση οδηγία της Επιτροπής. Δεν θα πρέπει να ξεχνάμε την κοινοτική στρατηγική για το εμπόριο, την οποία συζητάμε ελάχιστα. Όσον αφορά την ενεργειακή πολιτική της Ευρωπαϊκής Ένωσης, όλοι γνωρίζουμε ποιοι είναι οι κίνδυνοι των αναπτυσσομένων χωρών όσον αφορά τις πρώτες για την παραγωγή βιοκαυσίμων. Μετακίνηση πληθυσμών, ε, μείωση των εδαφών που χρησιμοποιούνται για τις ε, διατροφικές καλλιέργειες κλπ. Είναι κατεπήγον λοιπόν η εισηγήτρια να ζητήσει από την Κομισιόν αξιόπιστα στοιχεία για τις έμεσες συνέπειες της καλλιέργειας βιοκαυσίμων. Όσον αφορά τις μεταναστευτικές ροές, με ικανοποίηση διαπιστώνω ότι η εισηγήτρια συμμερίζεται το φόβο μου ότι η υλοποίηση της μπλε κάρτας για τους ε, μετανάστες δεν βοηθάει τους ε, μετανάστες ε, που προέρχονται από αναπτυσσόμενες χώρες και που έχουν προσόντα. Όσον αφορά δε τις εξαγωγές όπλων, πρέπει να υπάρχει κάποιος ε, περιοριστικό, ένα περιοριστικό πλαίσιο. Θέλω να, απογοήτε, να εκφράσω την απογοήτευσή μου όπως και ο κύριος Γκέρενς, που βλέπω ότι μόνο δύο άλλες κοινοβουλευτικές επιτροπές θα γνωμοδοτήσουν για αυτή τη σημαντική έκθεση. Λόγω της εξωτερικής ε, επιρροής της ε, εμπορικής πολιτικής, η Ήγκρα και η Ίντε δυστυχώς δεν συμμετέχουν στην εργασία αυτή. Παρά τα θα κάνουμε ό,τι μπορούμε για να συνεργαστούμε στενά με τη μόνιμη συγγήτρια, ώστε να μπορέσει το Κοινοβούλιο να εκφράσει ένα ισχυρό μήνυμα προς το Συμβούλιο και προς την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Σας ευχαριστώ. Taylor, the... Κύριε Τέιλορ, έχετε το λόγο. Oh, well, thanks very much, Chair. Ευχαριστώ πολύ, Πρόεδρε. Πολύ καλή έκθεση. Ευχαριστούμε πολύ. το θέμα της πολιτικής συνοχής για την ανάπτυξη είναι τόσο σημαντικό που πραγματικά πιστεύουμε ότι θα έπρεπε να είναι μια γενικότερη στρατηγική στα πλαίσια όλων των, των επιτροπών του Κοινοβουλίου να εργάζονται στα πλαίσια μια συνεκτικότητας. Μέχρι πρόσφατα ήμουν μέλος της Επιτροπής Διεθνούς Εμπορίου, όπου συζητούν τα θέματα εμπορίου και δεν ε, ξέφευγαν πολύ από αυτό. Παραδείγματο χάρη, η Επιτροπή Εμπορίου συζητούσε τις αναθεωρήσεις των GSP, τον GSP. Απογοητεύτηκα ιδιαίτερα που διαπίστωσα ότι ε, χρησιμοποιήθηκε ως μοναδικός καθοριστικός παράγοντας για το που θα πρέπει να το GSP το μέσο ανώτερο εισόδημα πολλών χωρών. Δεν υπάρχει ευαισθησία, δεν συζητώνται τα θέματα της, το πόσο ευάλωτες είναι χώρες και οικονομίες. Οι οικονομίες έχουν, ε, ε, ε, γίνει εξαρτημένες από πολύ λίγα ζητήματα. Και μόνο αυτό το παράδειγμα έδειξε ότι η πρόοδος μπορεί να αντιβαίνει τους αναπτυξιακούς στόχους της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Γι' αυτό ακριβώς είναι σημαντική η συνοχή της αναπτυξιακής πολιτικής. Θέλω να συνεργαστώ με την εισηγήτρια και τους σκιώδες και με τις άλλες επιτροπές επ' αυτού. Επειδή απλά και μόνο χρειαζόμαστε μια ευρύτερη εικόνα και εδώ έχουμε μια ευρύτερη εικόνα που θα μας βοηθήσει το έργο αυτής της έκθεσης είναι πολύ θετικό, είναι ιδιαίτερα θετικά κάποια στοιχεία του, όπως η ανάγκη να δοθεί περισσότερη προσοχή στην κλιματική αλλαγή και στις συνέργειες που ε, υπάρχουν σχετικά. Παράγραφοι 17 και 18 ζητούν να αξιολογηθεί ο ρόλος, η σημασία και η δυνατότητα αλλά και οι κίνδυνοι που προκύπτουν από τα βιοκαύσιμα. Δεν θα πω πολλά περισσότερα κυρία Πρόεδρε. Προσβλέπω στην ε, δουλειά για την έκθεση αυτή γιατί προσφέρει πολλές δυνατότητες. Ευχαριστώ. Merci. Ε, Ευχαριστώ. Παίρνω και εγώ τον λόγο για να ευχαριστήσω την εισηγήτρια για τη δουλειά της και για να πω ότι προσωπικά θεωρώ ότι είναι μια ευκαιρία να εισάγουμε κάτι, την ιδέα αυτή πιο συγκεκριμένα. Δηλαδή δεν γνωρίζουμε σήμερα εμείς τις αντιφάσεις που υπήρξαν μεταξύ της πολιτικής αλίας και της πολιτικής ανάπτυξης, Φερρυπίν. Δεν μπορούμε να, το να τις υπογραμμίσουμε αυτές με λιγότερο πολιτικά ορθό τρόπο όπως και η αγροτική μας πολιτική. Εδώ γνωρίζουμε πράγματα που θα μπορούσαμε να υπενθυμίσουμε επ' ευκαιρία της έκθεσης αυτής. Να υπενθυμίσουμε ότι ο λευτικός μας στόλος στην Δυτική Αφρική Φερρυπίν έχει κάνει πράγματα που δεν θα θέλαμε να επαναληφθούν που δεν θα έπρεπε να επαναληφθούν. Δεν αρκεί ίσως να πούμε ότι πρέπει να, να έχουμε υψηλό επίπεδο ανάληψη ευθύνη. Ξέρω ότι αυτά είναι αμφιλεγόμενα πράγματα, αλλά έχουν γίνει επιστημονικές μελέτες σχετικά και ίσως θα έπρεπε να κάνουμε και μια αναφορά στις επιστημονικές μελέτες που δείχνουν τις αντιφάσεις αυτές ε, που έχουν παρατηρηθεί μέχρι τούδε στις διάφορες της Ένωσης. Αυτά και τώρα θα δώσω το λόγο στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή, στην κυρία Φρανσουάς Μωρό. Θέλετε το λόγο. Ευχαριστώ. Καταρχήν, να υπογραμμίσω τη σημασία που έχει η έκθεσή σας στην Επιτροπή Ανάπτυξης. Είναι η πρώτη φορά που το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο από τότε που η Ευρωπαϊκή Επιτροπή όρισε μια ατζέντα, ένα συγκεκριμένο πρόγραμμα για αυτή την ανάπτυξη. Είναι η πρώτη φορά λοιπόν που το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο μας παρουσιάζει μια έκθεση σφαιρική θα λέγαμε σε θέματα συνοχής που βλέπει όλες τις πτυχές, τη κλίμα, ευρωτική παραγωγή και θεωρούμε είναι πραγματικά ένα στάδιο πάρα πολύ σημαντικό του λεχθέντος, όπως υπογράμμισαν πολλοί προαλαλήσαντες, όταν δουλεύει κανείς με τη συνοχή, υπάρχουν και άλλες ε, επιτροπές και άλλες υπηρεσίες που δουλεύουν για την ανάπτυξη και ξέρουμε πολύ καλά έχουμε ένα, ε, μια, ένα, μια ομάδα η οποία δουλεύει και συνεργάζεται με διαφορετικές υπηρεσίες είναι πολλές φορές δύσκολα να εξηγήσει κανείς κάποιες πτυχές και φυσικά ακόμα δυσκολέτερα να καταλήγει κανείς σε συγκεκριμένα αποτελέσματα. Θα προσπαθήσουμε να κάνουμε στα πάντα και συμφωνώ με αυτά που λένε οι προαλήσοντες ότι είναι σημαντικό και ότι θα πρέπει και άλλες επιτροπές του Κοινοβουλίου να ενταχθούν και να συνεργαστούν για αυτή την έκθεση. Ένα άλλο σημείο που θα ήθελα να θίξω είναι να διασφαλίσω στην Επιτροπή σας ότι από την Επιτροπή την Ευρωπαϊκή δεν υπάρχει πρόθεση να μειωθούν οι προσπάθειες που καταβάλλονται για αυτή την πολιτική και πραγματικά υπάρχει θέληση ίσως ο τρόπος να μην ήταν σωστός αλλά πραγματικά ειλικνά θα ήθελα να επιμείνω ότι ε, λειτουργούμε στα πλαίσια της συνθήκης, ε, τηρούμε τις δεσμεύσεις του 2005 για θέματα που έχουν να κάνουν με την ανάπτυξη και του 2009 και όπως επιθύμησαν και πολλοί υπάρχουν και άλλες, ε, άλλα μέσα όπως το άρθρο 12 για το Κοτονού υπάρχει και όπως ανέφερα η, ομάδα ανάμεσα στις διαφορετικές υπηρεσίες της Επιτροπής και αυτό που κάνουμε είναι να προσπαθούμε να πετύχουμε μια ανάλυση για ένα συγκεκριμένο πρόγραμμα για τις επόμενες μήνες να, να εντοπίσουμε, να προσδιορίσουμε κάποιες ε, ε αποφάσεις, κάποιες ε, προτεραιότητες και να δούμε τι μπορούμε να κάνουμε εν δυνάμει στους στόχους που έχουν οριστεί. Και θα συνεχίσουμε ενεργητικά ούτως ώστε ε, να λάβουν υπόψη οι μελλοντικές ε, αποφάσεις των επιτρόπων όλες αυτές τις πτυχές. Σε, τώρα για το σχέδιο της εκθεσής σας που έχετε, αν μου επιτρέπετε να αφήσω το συνάδελφό μου να κάνει και αυτός κάποια σχόλια σε, σχέση με, τις, με άλλες υπηρεσίες. Εγώ αυτό που θα ήθελα να πω ότι είναι σημαντικό το θέμα της κατάρτισης και προσπαθούμε σε ευρωπαϊκό επίπεδο να προετοιμάσουμε ένα πρόγραμμα κατάρτισης και να διασφαλίσουμε πόρους, κονδύλια για αυτό το πρόγραμμα. Είναι σημαντικό να επεξηγήσουμε αυτό το θέμα, διότι είναι σημαντικό για το πρόγραμμα συνοχής. Επίσης, να πω ότι έχουμε κινητοποιήσει την ομάδα μας που ανέφερα στην Επιτροπή. Μπορούμε να περάσουμε κάποια, να περάσουμε τα σχόλια, να σας ενημερώσουμε για κάθε θέμα. Αυτό που ελέγχθη για την αγροτική πολιτική και το εμπόριο τώρα. Για το εμπόριο. Έχουν γίνει δύο διαφορετικές ανακοινώσεις, αλλά δεν νομίζω ότι αυτό αποτελεί αυτό καθ' αυτό ένα πρόβλημα διότι καταρχήν έγινε μια ανακοίνωση για την ανάπτυξη και το εμπόριο και αυτό μας επέτρεψε να βαθύνουμε τη συζήτηση με τις ε, συναδέλφους μας στη Γενική Διεύθυνση για το Εμπόριο και να προβλεφθούν κάποιες συγκεκριμένες δράσεις. Δεν θα μπορούσαμε αυτό να το κάνουμε με μια γενική ανακοίνωση, καταλαβαίνετε. Αυτό είναι ένας περιορισμός για να μπορέσει να κάνει μια ουσιαστική συζήτηση. Για τις χώρες ΑΚΕ, και εδώ πέρα έχουμε θέματα τα οποία θα σας ε, τα ανακοινώσουμε αν το θέλετε. Για την αγροτική πολιτική τώρα. Αυτό που διαπιστώνει κανείς είναι ότι η κοινή αγροτική πολιτική έχει εξελιχθεί ουσιαστικά από το 2003-2004. Οι προτάσεις της Επιτροπής που έγιναν για την επόμενη δημοσιονομική περίοδο ε, εντάσσουν σε αυτά τη διάσταση που εμεί θέλουμε και η οποία είναι ικανοποιητική το πράγμα αυτό και στις συζητήσεις που έχουμε με τον συνάδελφό μου, με την αρμόδια γενική διεύθυνση. Θεωρούμε τα θέματα που χωρούν προς τη σωστή κατεύθυνση όσον αφορά και τις εξαγωγές και αντιμετωπίζουμε και το θέμα του ώστε να μην γίνεται επικάλυψη όσον αφορά τις, ε, τη βοήθεια. η κοινή αγροτική πολιτική, η σημερινή και η μελλοντική, λαμβάνει πάντα πολύ υπόψη το θέμα της συνοχής. Και αυτό πρέπει να το υπογραμμίσουμε στα πλαίσια μιας θετικής προοπτικής. Ευχαριστώ, Πρόεδρος. Υπάρχει κάποιος άλλος από την Επέτροπη που θα επιθυμούσε να πάρει το λόγο για το θέμα της ε, συνοχής των πολιτικών. Όχι. Οπότε, να δώσω το λόγο για τις υπηρεσίες εξωτερικών δράσεων στον Ούλα Σιρστρέμ. Θα δώσω το λόγο. Ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε. Θέλω να ευχαριστήσω την Επιτροπή σας αλλά και τη Φρανσουάς για τα καλά της λόγια. Να ευχαριστήσω και την εισηγήτρια. Πράγματι, είναι ένα εξαιρετικό ε, εξαιρετικά σημαντικό θέμα αυτό, το, ε, η συνοχή της αναπτυξιακής πολιτικής και μπορέσατε όλοι να, μπόρεσε η συγγήτρια να συμπεριλάβει τόσο πολλά θέματα σε τόσο σύντομο κείμενο. Πολύ σωστά είπε επίσης ότι είναι ένα πολύ περίπλοκα τεχνικό ένα πολύ περίπλοκο ζήτημα από την τεχνική σκοπιά αλλά και από την πολιτική σκοπιά. Συμφωνώ απολύτως με αυτά που είπε η Φρανσουάζ κατά τα λοιπά. Ενδεχομένως κάποιες τεχνικές παρατηρήσεις έχουμε να κάνουμε για το κείμενο. Σε αυτό το στάδιο θα ήθελα μόνο να σχολιάσω την πέμπτη παράγραφο της έκθεσης και να πω το εξής. Τονίζεται ότι έχει σημαντικό ρόλο η υπατή εκπρόσωπος μέσω της εξωτερικής δράσης, μέσω της υπηρεσίας για τις εξωτερικές δράσεις. Εμείς θεωρούμε ότι το πιο ο πιο σημαντικός ρόλος για την ύπατη εκπρόσωπο είναι το γεγονός ότι είναι αντιπρόεδρος και της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και έτσι διασφαλίζεται η συνοχή της πολιτικής που έχουμε ως Ευρωπαϊκή Ένωση για την ανάπτυξη. Είναι σημαντικό κατά την άποψή μου. Αλλά βεβαίως θα επανέλθω αργότερα με περισσότερα σχόλια. Ευχαριστώ. Η Πρόεδρος, ευχαριστώ πολύ. Να δώσω ξανά το λόγο στην κυρία Γιάστραμ για να κάνει τις καταληκτικές παρατηρήσεις. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Ευχαριστώ τους συναδέλφους που ε, παρενέβησαν και ευχαριστώ για τις προτάσεις του. Πολλές είναι ιδιαίτερα ενδιαφέρουσες, ιδιαίτερα του Γκέρεν ότι πρέπει να υπογραμμίσουμε και να δείξουμε τη σημασία ορισμένων τομέων. Υπάρχει το θέμα του συντονισμού ανάμεσα στις διάφορες επιτροπές και με αυτόν τον τρόπο μπορεί να δημιουργήσει κανείς ίσως μια αιτήσια έκθεση. Να έχει κανείς μια γενική έκθεση και μετά κάποια ε, εξειδικευμένη. Αυτό θα μπορούσε ίσως να προκαλέσει και το ενδιαφέρον των άλλων επιτροπών. Θα ενδιαφερόντουσαν, θα θεωρούσαν ότι έχουν λόγο, θα παίρναν θέση και θα μπορούσαν να συντάξουν νομοδοτήσει για το ΑΒ θέμα. Είναι σημαντικό θέμα το έχει εξάλλου δείξει η ε, συζήτηση. Στη συνάντηση που είχε γίνει με τις χώρες ΑΚΕ είχε θυχτεί το θέμα λέγοντας ότι εμείς θεωρούμε ότι θα πρέπει και οι χώρες ΑΚΕ να προβληματιστούν πάνω στα θέματα στα οποία μπορούμε να αντιμετωπίσουμε στα πλαίσια διαλόγου είναι κάτι που έχει να κάνει με δύο μέρη. Θα μπορούσαμε να μιλήσουμε ενδεχομένω και για την αλληλεία ακόμα. Είναι ένα θέμα το οποίο πραγματικά πρέπει να προβληματίζει. Χαίρομαι με αυτά που είπε η Επιτροπή όσον αφορά τις προοπτικές. Θα υπάρχει το, το Σεπτέμβριο θα υπάρξει ψηφοφορία στο Κοινοβούλιο και θα μπορούσαμε να ενημερωθούμε ευρετέρω για το γενικότερο διάρμα. Ευχαριστώ. Κατάθεση τροπολογιών προθεσμία είναι 19 Ιουλίου και θα ψηφίσουμε για αυτή την έκθεση ε, το Σεπτέμβριο. 19 Ιουλίου, μεσημέρι, 12 η ώρα για τις απολογίες. Προθεσμία κατάθεση τροπολογιών εγγών. Λοιπόν. Τώρα περνάμε στο σημείο 15 η Συμφωνία Σύνδεσης ανάμεσα στην Ευρωπαϊκή Ένωση και τα κράτη-μέλη της από τη μία και την Κεντρική Αμερική από την άλλη. Λοιπόν, είναι νομοθετική γνωμοδότηση για τη συμφωνία σύνδεσης και από την άλλη έχουμε μια μη νομοθετική γνωμοδότηση που έχει να κάνει με προτάσεις στα πλαίσια θεμάτων τα οποία σε μεταβατικό στάδιο και στο οποίο έχουμε εισηγητή τον Σάλα Φράγκα. Η Ευρωπαϊκή Ένωση και η Κεντρική Αμερική το Μάιο του 2010 ολοκλήρωσαν τις συνομιλίες για μια συμφωνία σύνδεσης στηριζόμενη σε τρεις πυλώνες, διάλογος πολιτικό, συνεργασία και εμπόριο. για να περάσει να έχει νομική βάση θα πρέπει αυτή η συμφωνία να εγκριθεί, επικυρωθεί τόσο από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο όσο και από τα κοινοβούλια των χωρών μελών. Αυτή η νέα συμφωνία θέλει να ενισχύσει την πολιτική και οικονομική σταθερότητα στις χώρες της Κεντρικής Αμερικής και να τι ενισχύσει να οδηγηθούν σε μια βιώσιμη ανάπτυξη σε περιφερειακό επίπεδο. Η συγγήτρια εκεί για τις διονομοδοτήσεις είναι η κυρία Γκρέζ, η οποία δεν είναι εδώ, η οποία όμως μου ανέθεσε να σας διαβάσω την γνωμοδότησή της. Λοιπόν, θα είμαι η φωνή της Κατερίν Κρέζ, που είναι η, γνω... η συγγνώμη, αυτών των δύο γνωμοδότησεων. Αγαπητοί συνάδελφοι, η, η Κατερίν Κρέζ από τους Πράσινους είναι αυτή που κάνει την γνωμοδότηση για τη Συμφωνία Σύνδεσης με τις Κεντρική Αμερική. Και συζητήσει γνώμη που θα λείπει. Γίνεται μια ανταλλαγή απόψεων για δύο διαφορετικές γνωμοδοτήσεις, αλλά που είναι σχετικές. Η μία είναι η έγκριση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου για την Συμφωνία Σύνδεσης με την Κεντρική Αμερική και η δεύτερη αφορά την άποψη της Επιτροπής Ανάπτυξης για την ενδιάμεση έκθεση της Επιτροπής Εξωτερικών Σχέσεων για την σχέση για την ε, ε, Συμφωνία ε, Σύνδεσης. Η συμφωνία αυτή στηρίζεται σε τρεις πυλώνες, τον πολιτικό διάλογο, τη συνεργασία και την εμπορική συμφωνία. Δεδομένου ότι το εμπόριο είναι σημαντικό στοιχείο της βιώσιμης ανάπτυξης, η ομάδα των Πρασίνων θεωρεί ότι η εμπορική συμφωνία δεν πληρεί τους απαραίτητους όρους. Δεν αποδεικνύει κατ' ουδένα τρόπο ότι θα υπάρξουν ωφέλη για τον πληθυσμό και δεν λαμβάνει υπόψη τις ασυμμετρίες που υφίστανται σε σχέση με τα επίπεδα ανάπτυξης. Αν οι χώρες Κεντρικής Αμερικής έχουν υψηλά επίπεδα φτώχειας, το 50% του πληθυσμού ζει σε κατάσταση φτώχειας, τα πλεονεκτήματα που θα μπορέσουν να ε, έχουν από την προτιμησιακή αυτή ε, συμφωνία ε, εξαρτώνται από το γεγονός ότι οι περισσότερες εξαγωγές της Κεντρικής Αμερικής ήδη έχουν πρόσβαση ε, στις ε, ε, αγορές της Ευρωπαϊκής Ένωσης με το καθεστώς ΣΥΓΜΑΓΑΜΑΠΗ+. Η εκτίμηση των επιπτώσεων για τη βιωσιμότητα αφορά κυρίως τους τομείς που αφορούν τα σημαντικότερα μέρη της οικονομίας αυτών των χωρών. Έτσι λοιπόν η συμφωνία μάλλον θα ενισχύσει την ε, αυξημένη εξάρτηση από εξαγωγές πρωτογενών γεωργικών προϊόντων. Με την σύναψη συμφωνιών ΠΟΕ-ΣΥΝ σχετικά με τις δημόσιες συμβάσεις, την απελευθέρωση υπηρεσιών και τα δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας, η παρούσα συμφωνία με τις χώρες Κεντρικής Αμερικής περιορίζει το πεδίο άσκησης πολιτικής τους ως προς τη δυνατότητα διαμόρφωσης της δικής τους αναπτυξιακής στρατηγικής ή ως προς τη δυνατότητα εκπόνησης συγκεκριμένων μέτρων που θα εγγυώνται ότι οι επενδύσεις αποβαίνουν προς όφελος των φτωχών και των πλέον ευάλωτων. Η γνώμη τη συντάκτη παρούση είναι ότι η συμφωνία πάσχει από σειρά σοβαρών μειονεκτημάτων που άπτονται ε, θεμάτων ε, δικαιωμάτων εργασιακών κτλ μπορεί να οδηγήσει σε μείωση της ε, παραγωγής ε, τροφίμων και την μετακίνηση, στη μετακίνηση πληθυσμών. Η συμφωνία ε, πάσχει από σοβαρά κενά όσον αφορά τα ανθρώπινα δικαιώματα, τα, τις συνθήκες εργασίας και τα θέματα περιβάλλοντος και βιώσιμης ανάπτυξης. Αν θέλουμε παρότι η ενσωμάτωση ρήτρας ανθρωπίνων δικαιωμάτων είναι ευπρόσδεκτη, παρά τα αυτά πάσχει από σοβαρά μειονεκτήματα. Δεν υπάρχει συγκεκριμένο τμήμα αφιερωμένο στην επιτήρηση της συμμόρφωσης με αυτή την υποχρέωση. Η υποχρεωτική εφαρμογή της Ρήτρας δεν υπόκειται στο μηχανισμό επίλυσης διαφορών και παραλείπει οποιαδήποτε σημαντική αναφορά στην εταιρική κοινωνική ευθύνη και στη σύμβαση σε 169 του ΔΟΕ, της ΔΟΕ. Για όλους αυτούς τους λόγους η Επιτροπή Ανάπτυξης θα πρέπει να ζητήσει από την αρμόδια επί της ουσίας Επιτροπή Εξωτερικών Σχέσεων να ζητήσει από το Κοινοβούλιο να αρνηθεί την έγκριση αυτής της συμφωνίας και να συμπεριλάβει αυτές τις ανησυχίες της στην ενδιάμεση εκθεσή της. Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο θα πρέπει να ε, να, ψηφίσει την μη ισόρροπη αυτή έκθεση το επόμενο φθινόπωρο. Ως εισηγήτρια της Επιτροπής Ανάπτυξης ζητώ από όλους τους συναδέλφους να απορρίψουν την ε, έκθεση. Για συμπληρωματικές πληροφορίες, στις 29 Ιουνίου η συμφωνία της σύνδεσης υπογράφηκε στην Τέκη Συγκάλπα, την πρωτεύουσα των, της Ονδούρας. Η υπογραφή αυτή έγινε 300 μέρες ακριβώς μετά το ε, ε, πραξικόπημα του 2009 που έγινε στην Ονδούρα. Υπάρχει θέμα σοβαρό ε, ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Παρά τα αυτά, η Επιτροπή έστειλε ένα πολύ αρνητικό μήνυμα θέτοντας το εμπόριο πάνω από τα ανθρώπινα δικαιώματα. Η συμφωνία αυτή περιέχει ένα κεφάλαιο ελεύθερων ανταλλαγών και δεν είναι καθόλου κατάλληλη στιγμή να υπογραφεί 300 ημέρες μετά το πραξικόπημα στην Ονδούρα που ε, αφήνει τιμώρητες ε, πολλές πολιτικές δολοφονίες. Η Ευρωπαϊκή Ένωση μοιάζει να επιδιώκει μόνο ε, με τα, με επιμονή στο μοντέλο αυτό ανάπτυξής της η συμφωνία αυτή σύνδεσης θα είναι εξαιρετικά επωφελής για τις ευρωπαϊκές επιχειρήσεις γιατί θα τους ανοίξει πρόσβαση στον τομέα τηλεπικοινωνιών, στον τουρισμό, στο νερό, στην ενέργεια και στις δημόσιες προμήθειες. Αντιθέτως, δεν θα βελτιώσει τις συνθήκες ζωής του τοπικού πληθυσμού. Τα λόγο έχουν πλέον τα μέλη της Επιτροπής. Ο κύριος Κόρτες Λάστρα έχει ζητήσει το λόγο. Παρακαλώ. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Αντιθέτως, εγώ πιστεύω ότι πρέπει να ε, είμαστε ικανοποιημένοι με τη Συμφωνία Σύνδεσης Κεντρικής Αμερικής και Ευρωπαϊκής Ένωσης. Είναι η πρώτη συμφωνία σύνδεσης που υπογράφεται μεταξύ δύο διαφορετικών περιοχών, δύο διαφορετικών περιφερειών και είναι διαφοροποιημένη η συμφωνία αυτή σε σχέση με τις αποκλειστικά εμπορικές συμφωνίες. Δεν είναι μια συνθήκη ελεύθερων συναλλαγών, είναι μια πραγματική συμφωνία η οποία θέτει σε ισότιμη βάση τις δύο περιφέρειες αυτές. Ως εκ τούτου δίνεται η δυνατότητα σε αμφότερα μέρη να έχουν ε, πολιτική παρέμβαση σε θέματα δημοκρατίας και ανθρωπίνων δικαιωμάτων και δεν απλά ε, γίνεται μια πολύ ισχυρή επιχειρηματολογία υπέρ των ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Επιτρέπεται η υιοθέτηση μέτρων όταν καταστρατηγούνται αυτά τα ανθρώπινα δικαιώματα που μπορούν να φτάσουν και μέχρι την αναστολή της εφαρμογής της συμφωνίας. Προβλέπεται δημιουργία σύσταση κοινοβουλευτικής επιτροπής και δίδεται όθηση στις εργασίες ε, και τις συστάσεις ε, του Πάρλα Σεν είναι πολύ σημαντικό το ότι η συμφωνία λαμβάνει υπόψη της τις ασυμμετρίες που υπάρχουν στην περιοχή εκεί. Και μόνο με αυτόν τον τρόπο μπορούμε να οδηγηθούμε σε περιφερειακή ολοκλήρωση και να πετύχουμε πραγματικά αυτή την περιφερειακή ολοκλήρωση. Η Κεντρική Αμερική ε, μαζί με τη Λατινική Αμερική γενικότερα, είναι μια περιοχή με τις μεγαλύτερες ανισότητες στον κόσμο. Και γι' αυτό εμείς εδώ δίνουμε έμφαση στον αγώνα κατά των ανισοτήτων. Συμπεραίνω λέγοντας ότι αυτή η επιτροπή, η συμβουλευτική και διαβούλευση για όλα αυτά τα θέματα είναι εξαιρετικά σημαντική. Το πιο σημαντικό όμως είναι να εφαρμοστούν στην πράξη οι συστάσεις της Επιτροπής. Πρέπει να διπλασιάσουμε τις προσπάθειές μας ώστε να έχουμε αποτελεσματική συμμετοχή της οργανωμένης ε, ε, κοινωνίας των πολιτών. Ευχαριστώ πολύ. Η Πρόεδρος. Ευχαριστώ. Ο κύριο Φίσας Εξέλα. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Και εγώ θα ήθελα να ευχαριστήσω την κυρία Γκρέσ για τη δουλειά που έχει κάνει κατά τη σύνταξη αυτών των δύο ε, γνωμοδοτήσεων, παρόλο που ενδεχομένως τα συμπεράσματά μας αποκλίνουν. Αυτή τη στιγμή ε, δουλεύουμε πάνω στις τροπολογίες για τη μη νομοθετική γνωμοδότηση και ελπίζουμε ότι με τις τροπολογίες που θα καταθέσουμε πράγματι θα βελτιωθεί το κείμενο και πράγματι θα διασκεδαστούν κάποιες από τις ανησυχίες που έχει η συγγήτρια κυρία Κατρίν Γκρέτζ ως προς τα θέματα αυτά. Όπως αναφέρει και ο κύριος Αλαφράγκα, ο εισηγητής της σχετικής έκθεσης από την Επιτροπή Εξωτερικών Υποθέσεων, θέλω και εγώ να επισημάνω ότι η Συμφωνία Σύνδεσης μεταξύ ΕΕ και Κεντρικής Αμερικής πράγματι συμβάλλει στην επίτευξη των στόχων της εξωτερικής πολιτικής της Ευρωπαϊκής Ένωσης και ενισχύει την ε, περιφερειακή ολοκλήρωση, όπως άλλωστε το είπε και ο κύριος Κορτές που μόλις τώρα πήρε το λόγο και όπως άλλωστε είπε ότι είναι η πρώτη συμφωνία τέτοιου είδους που συνάπτει η Ευρωπαϊκή Ένωση με τα, ε, χώρες της περιοχής αυτής. Σε αυτό το πλαίσιο λοιπόν θέλω να επισημάνω ότι η συμφωνία αυτή δίνει προτεραιότητα στα κοινωνικά ζητήματα. Ότι αυτός δηλαδή είναι ο στόχος της περιφερειακής πολιτικής. Και βασική προτεραιότητα είναι η μείωση του ποσοστού της φτώχειας, της ανισότητας, του κοινωνικού αποκλεισμού και ε, οποιασδήποτε διάκριση τέτοιου είδους. Γίνεται λόγος για τα ανθρώπινα δικαιώματα επίσης και θεωρούμε εμείς ότι ε, η συμφωνία αυτή επιμένει ιδιαίτερο στην εφαρμογή και στην τήρηση των δημοκρατικών αρχών, στο σεβασμό του κράτους δικαίου και ε, πιστεύουμε ότι όλα αυτά είναι εξαιρετικά θετικά. Με τη συμφωνία αυτή μπορεί να γίνουν ευρωπαϊκές επενδύσεις, παρόλο που διανύουμε κρίση, μια περίοδο κρίση στην Ευρώπη αυτή τη στιγμή. Θα γίνουν επενδύσεις στην περιοχή από πλευράς Ευρώπη και αυτό θα έχει πολύ θετικό αντίκτυπο στην τοπική κοινωνία. Όσες περισσότερες επενδύσεις γίνονται, τόσο περισσότερη απασχόληση θα υπάρχει εκεί στην περιφέρεια, στην περιφέρεια της Κεντρικής Αμερικής. Δεν βλέπω λοιπόν να υπάρχει καμία σύγκρουση μεταξύ του εμπορικού σκέλου και του ε, ανθρώπινου, αν θέλετε, σκέλους. Αντιθέτως, Κατά τα λοιπά, ως πολιτική ομάδα είμαστε στη διάθεσή σα να υποβάλουμε τροπολογίε και να εργαστούμε για την βελτίωση του κειμένου. Ευχαριστώ πολύ. Η Πρόεδρος, ο κύριος Γκέρανς, έχει το λόγο. Παρακαλώ. Ευχαριστώ κυρία Πρόεδρε. Η κυρία Γκρέζ στις γνωμοδοτήσεις της αναλύει επισταμένος τον αντίκτυπο της εμπορικής αυτής συμφωνίας στις χώρες της Κεντρικής Αμερικής. Αναφέρεται σε προφανείς αλήθειες. Το εμπόριο δημιουργεί πλούτο, αλλά δεν εγγυάται την σωστή κατανομή αυτού του πλούτου. Και αυτό αληθεύει το έχουμε διαπιστώσει όταν συζητούσαμε τα θέματα της διαφοροποίησης. Εν πάση περιπτώσει, αναρωτιέμαι, τα μέσα που προτείνει η συγκήτρια για την αποκατάσταση ε, ε της ε, ορθής τάξης πραγμάτων είναι πράγματι τα σωστά. Έχει απόλυτο δίκιο όσον αφορά στα ανθρώπινα δικαιώματα. Ε, το σκέλος του κειμένου εκεί πράγματι επιδέχεται βελτιώσεων. Αναλύει τον αντίκτυπο έχει το εμπόριο στην παραγωγή την εγχώρια των χωρών αυτών, δεν σφάλει σε αυτά που λέει, πράγματι ελοχεύει ο κίνδυνος οι χώρες αυτές να εξαρτώνται άμεσα από τις εξαγωγές των προϊόντων τους. Και τελικά να ε, αυξάνονται οι κίνδυνοι για τους πληθυσμούς τους. Για να αποκαταστήσουμε λοιπόν ε, το τοπίο ε, μπορούμε να ακολουθήσουμε διαφορετικές άγουσες. Η κυρία Γκρέζ μας καλεί να απορρίψουμε τη συμφωνία αυτή. Ε, αυτό είναι όμως μία και έξω. Είναι κάτι που γίνεται μία και έξω. Ε, μπορεί όντως να πούμε ότι η Επιτροπή πιστεί στους στόχους της για τη βιώσιμη ανάπτυξη και για τη συνοχή των αναπτυξιακών πολιτικών καλεί το Κοινοβούλιο να απορρίψει τη συμφωνία αυτής σύνδεσης. Ε, όπως ε, είπα και προηγουμένως, είναι κάτι που γίνεται εφάπαξ. Άρα πώς θα μας μείνουν ε, εργαλεία μετά για να ασκήσουμε πίεση στις χώρες αυτές. Άπαξ και απορριφθεί, απορρίφθηκε. Μπορούμε βέβαια από την άλλη να δεχθούμε τη συμφωνία και να δούμε ποια είναι τα εργαλεία που έχουμε στη διάθεσή μας, τα μέσα. Πρώτον, ο πολιτικός διάλογος. Δεν ταυτίζεται βέβαια με ένα μέσο άσκησης έντονης Ωστόσο, εκεί μπορούμε να ε, χειριστούμε αυτό το μέσο για να ε, πιέσουμε αυτές τις χώρες. Έχουμε και την αρχή της διαφοροποίησης της βοήθειας. Δεν ξέρω σε ποιο βαθμό θα μπορούσε να εφαρμοστεί στις χώρες της Κεντρικής Αμερικής. Ωστόσο, χώρες που φτάνουν σε ένα συγκεκριμένο επίπεδο παραγωγής ε, πλούτων μπορούν να βγουν ενδεχομένω από τον κατάλογο δικαιούχων ε, και αντιστοίχως. Ε, προτείνω να αξιοποιήσουμε περισσότερο αυτά τα εργαλεία. Εγώ προτιμώ να παίξω με αυτά τα χαρτιά στο χέρι παρά να απορρίψω τη συμφωνία εξ αρχή. Καλό θα ήταν να μην στερηθούμε ε, τα μέσα δράσης μας. Και όπως και για άλλες συμφωνίες και για αυτή τη συμφωνία μπορούμε να αναρωτηθούμε το εξής είμαστε εμείς υπεύθυνοι για την εσωτερική τους πολιτική ή μήπως αυτές οι χώρες είναι υπεύθυνε για την εσωτερική τους πολιτική και για τον καθορισμό των προτεραιοτήτων του σε εσωτερικό επίπεδο. Δηλαδή ο διάλογος έχει και κάποια όρια. Μπορούμε βεβαίως και πρέπει να κάνουμε έναν επικοδομητικό επικοδομητικό διάλογο με τις χώρες αυτές, αλλά δεν μπορούμε τίποτα να τους επιβάλλουμε. Και αν εφαρμόζουμε τα ίδια πρότυπα παντού, τότε δεν θα ε, κάνουμε εμπορικέ συναλλαγές ε, ε, με κανέναν σχεδόν, όχι μόνο στην Κεντρική Αμερική, αλλά ούτε και στην Βόρεια Αμερική ή στην Ασία. Τα λέω όλα αυτά για να πω ότι συμμερίζομαι απολύτω τι ανησυχίε και τι διαπιστώσει τη κυρία Γκρέζε. Έχει απόλυτο δίκιο. Ωστόσο, δεν συμφωνώ με τα μέσα που μα προτείνει για την άρση αυτών των ανισοτήτων και των αδικιών. Ευχαριστώ. Το, το λόγο έχει τώρα η Κομισιόν. Όχι. Καταρχήν η κυρία Δολόρης Ρωμαίο. Thank you, Chairman. Ευχαριστώ κυρία Πρόεδρε. Θα αναφερθώ στην ρήτρα ανθρωπίνων δικαιωμάτων που πράγματι περιέχει συμφωνία σε σχέση με τη συμφωνία του 2003, η οποία έχει συναυθεί με την Κεντρική Αμερική, εδώ σήμερα συμπεριλαμβάνουμε τα κατάλληλα μέτρα για την περίπτωση της παραβίασης των βασικών στοιχείων της συμφωνίας, ένα από τα οποία είναι η ρήτρα ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Η, δικαιολογία που δίνει η συγγήτρια είναι ότι δεν υπάρχει μηχανισμός παρακολούθησης ε, για ε, να παρακολουθεί την εφαρμογή της ρήτρας αυτής. Θέλω να υπογραμμίσω ότι αυτή καθ' αυτή η συμφωνία ε, θεσπίζει ε, ένα πολύ ολοκληρωμένο θεσμικό πλαίσιο που ε, επιβλέπει την τήρηση των συμφωνιών από δύο πλευρές. Υπάρχει ένα Συμβούλιο Συμφωνής, μια Επιτροπή, μια μικρή Κοινοβουλευτική Επιτροπή όπου θα συμμετέχει και το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και επίσης ζητάμε από την Κοινωνία των Πολιτών να συμμετέχει και αυτή αυτή, δεδομένου ότι η συμφωνία δημιουργεί μια επιτροπή και συμφωνία των πολιτών και από τις δύο πλευρές. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Ευχαριστώ. Το ρόλο έχει τώρα η Ευρωπαϊκή Επιτροπή που εκπροσωπεί την κυρία Κόντσα Πλάτ Μελάντο. Ευχαριστώ κυρία Πρόεδρε. Θα προτιμούσαμε να πάρει το λόγο η Γενική Διεύθυνση Εμπορίου εκ μέρους της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και αν υπάρχουν άλλα θέματα σχετικά με την ανάπτυξη, τότε θα πάρω εγώ το λόγο. Πολύ ωραία. Δώμε το λόγο λοιπόν με διαφορετική σειρά στους εκπροσώπους της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Ευχαριστούμε για την ευκαιρία να συμμετέχουμε στη συζήτηση Φυσικά θα παρακολουθούμε με ενδιαφέρον τις εργασίες Επιτροπής Ανάπτυξης και θέλουμε να συμμετέχουμε σε αυτές. Θέλω απλώς να επισημάνω λίγα σημεία που αφορούν τη συμφωνία αυτή. Αλλά θέλω και να αντιδράσω σε ένα από τα δύο θέματα του σχεδίου γνωμοδότησης. Καταρχήν συμφωνώ απόλυτα με τα μέλη του Κοινοβουλίου που πήραν το λόγο και είπαν ότι το αποτέλεσμα είναι θετικό και για την Ευρωπαϊκή Ένωση και για την Κεντρική Αμερική. Εμείς από πλευράς Ευρωπαϊκής Ένωσης ε, ξέρουμε ότι για τις διαπραγματεύσεις στον πυλώνα του, του εμπορίου θέλαμε να πετύχουμε φιλόδοξα πράγματα, να επιτύχουμε κάτι θετικό για τις ε, ευρωπαίους εξαγωγείς προϊόντων και υπηρεσιών. Επιπλέον, υπάρχουν ε, ανοίγματα στην αγορά για τις χώρες Κεντρικής Αμερικής σε διάφορους τομείς και αν το συγκρίνουμε με τη δυνατότητα τις δυνατότητες που υπάρχουν στα πλαίσια της Συμφωνίας Γενικευμένων Προτιμήσεων, εδώ βλέπουμε ότι υπάρχουν πλεονεκτήματα για τη ζάχαρη, για τις μπανάνες, για το ρύζι και άλλα προϊόντα τα οποία δεν συμπεριλαμβάνονται στα πλαίσια του συστήματος γενικευμένων προτιμήσεων. Και φυσικά οι αγορές που έχουν κάνει μονομερείς παραχωρήσεις στο πλαίσιο αυτό για άλλα προϊόντα είναι σταθερές, δεν μπορούν να αλλάξουν και δεν υπόκεινται σε αβεβαιότητες όπως συνέβαινε στο σύστημα γενικευμένων προτιμήσεων όπου όταν επιτυγχάνονταν ένα συγκεκριμένο επίπεδο ευημερία έβγαιναν από το σύστημα. Τώρα, το δεύτερο στοιχείο που θέλω να υπογραμμίσω είναι ότι η συμφωνία αυτή ανταποκρίνεται σε μεγάλο βαθμό Στι πολιτικές προσεγγίσεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης ε, στη σχέση με τη Λατινική Αμερική Συμφωνία Σύνδεσης και επίσης συμπεριλαμβάνει ένα ισχυρό στοιχείο περιφερειακής ολοκλήρωσης που ε, έχουμε συμπεριλάβει σε όλες τις συμφωνίες μας με την Κεντρική Αμερική. Είναι η πρώτη ε, συμφωνία μεταξύ περιφερειών και στο στοιχείο εμπορίου υπάρχει ένα κεφάλαιο που οι χώρες Κεντρική Αμερικής δεσμεύονται να προχωρήσουν περισσότερο στον τομέα της οικονομικής ολοκλήρωσης. Και αυτό είναι σημαντικό στοιχείο. Ε, κάποιες ποσοστώσεις για το ρύζι, για τη ζάχαρη και για άλλα προϊόντα αποφασίζονται σε περιφερειακό επίπεδο. Δηλαδή η Κεντρική Αμερική θα πρέπει ε, στο εσωτερικό της να αποφασίσει για την κατανομή αυτών των ποσοστώσεων. Θεωρούμε ότι αυτό είναι σημαντικό στοιχείο για να μπορέσει να συνεργαστεί σε διάφορα θέματα η Κεντρική Αμερική και να ξεπεράσει την απλή πολιτική συνεργασία. Τώρα, ένα άλλο σημείο που θέλω να υπογραμμίσω διαπιστώσαμε μεγάλη πολιτική υποστήριξη από πλευράς ε, Κεντρικής Αμερικής προς τη συμφωνία αυτή. Το ένα επιχείρημα μας είναι ότι ακούστηκε ότι αυτή η συμφωνία δεν είναι καλή για την Κεντρική Αμερική, ότι επιβλήθηκε από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Αν δείτε τις ενδείξεις, τα μηνύματα και τις δηλώσεις των χωρών Κεντρικής Αμερικής ε, στην υπόθεση αυτή, θα δείτε ότι η κατάσταση είναι διαφορετική. Όπως γνωρίζετε έγινε ακρόαση στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, στην Επιτροπή ΙΤΑΣ, ΙΝΤΑΣ, την 30 Μαΐου αν δεν κάνω λάθος, κατά την οποία ακρόαση η Κεντρική Αμερική με την παρουσία διαφόρων υπουργών και πρέσβεων διατύπωσε ισχυρή πολιτική υποστήριξη προς τη συμφωνία αυτή. Η υπογραφή έγινε στις 29 Ιουνίου στην Ονδούρα, παρουσία και των έξι αρχηγών κρατών. Αυτό αποτελεί σοβαρότατο μήνυμα, σοβαρότατη ένδειξη υποστήριξης. Ε, με δύο λόγια, τα τελευταία δύο σημεία. Το σχέδιο σύστασης λέει ότι έχουμε ε, μια ρήτρα κοινωνικής εταιρικής ευθύνης στη συμφωνία. Αυτό δεν ισχύει. Περνάει στη συμφωνία λόγω του ότι συμπεριλαμβάνεται μια δέσμευση των πλευρών να διευκολύνουν την εταιρική κοινωνική ευθύνη και να συνεργαστούν περαιτέρω στον τομέα αυτό. Αν το συγκρίνεται με τους ε, δεσμευτικούς κανόνες που υπάρχουν για την εφαρμογή στα πλαίσια των συμβάσεων του ε, ΔΟΕ, πιστεύω ότι υποστηρίζεται η βελτίωση των συνθήκων εργασίας στην Κεντρική Αμερική και αποτελεί βήμα πρόοδου σε συνδυασμό με ε, σε σύγκριση με τις προηγούμενες συμφωνίες. Νομίζω λοιπόν ότι κάποια από τα θέματα αυτά ε, που ακούστηκαν και από την Επιτροπή Ανάπτυξης τα έχουμε αντιμετωπίσει. Τώρα θα πρέπει να συνεργαστούμε με την Κεντρική Αμερική ώστε να υλοποιηθούν όλα αυτά και αυτή θα είναι μία από τις δυσκολίες στο μέλλον. Ευχαριστώ. Euh, άλλοι που θα ήθελαν να πάρουν το λόγο από την Επιτροπή τουλάχιστον. Η κυρία Γκρές λοιπόν μέσω μου κλείνει το θέμα αυτό ε, λέγοντας ότι δεν έχουμε πιστεί λοιπόν με τα επιχείρηματά σας ε, θεωρούμε ότι αυτή η συμφωνία δεν είναι καλή υπάρχουν τόσα και τόσα προβλήματα, δολοφονίες, ε, ε, όσον αφορά δηλαδή το θέμα που έχει να κάνει με τα ανθρώπινα δικαιώματα, πραγματικά η κατάσταση είναι δραματική. Ε, είμαστε πολιτικοί, ξέρουμε πολύ καλά τη σημασία των συμβόλων για όσον αφορά την κατάσταση αυτή για τη συμφωνία που υπογράφει λοιπόν για την Ονδούρα. Ε, θα ήθελα να πω έχουμε μια κατάσταση όπου δεν υπάρχουν ωφέλη για τις χώρες τις οποίες αφορά τα κέρδη έχουν μεταφερθεί σε φορολογικούς παράδεισους. Ξέρουμε πολύ καλά ότι κάποιοι άλλοι έχουν κερδίσει, μέτοχοι. Έχουμε διάφορα προϊόντα όπως η Αυτό που διαπιστώνουμε ότι ε, οι τοπικοί πληθυσμοί δεν έχουν κερδίσει τίποτα και εκ μέρου της κυρίας Γκρέζ αυτό που ζητάω είναι να απορριφθεί αυτή εδώ η έκθεση. Κατάσταση τροπολογιών, προθεσμία, 3η Σεπτεμβρίου το, στις 12 το μεσημέρι. Και 18 Σεπτεμβρίου περνάει για ψηφοφορία στην Επιτροπή μας. Κλείνει η σημερινή συνεδρίαση. θα ξαναρχίσουμε στις 3. Συνεχίζοντας με άλλα θέματα εξίσου σημαντικά. Και πραγματικά ελπίζω να υπάρχει εκεί η παρουσία σας. Ευχαριστώ.